Nehmen Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να περάσετε καλά στις ε, διακοπές σας και να έχετε έρθει πίσω εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ανανεωμένοι. Σήμερα έχουμε την ε, ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό, τη συζήτηση για την αεροπορία, για την αεροκυκλοφορία. Ε, υπήρχαν τόσοι πολλοί ενδιαφερόμενοι που δημιουργήσαμε και ένα listening room και ελπίζω να βρούμε χρόνο και χώρο για όλους. Πρώτα απ' όλα για την ημερήσια διάταξη. Το σχέδιο ε, ημερήσιας διάταξης έχει εγκριθεί ή υπάρχουν αντιρρήσεις ενστάσεις. Όχι, από ό,τι βλέπω. Οπότε, συνεχίζουμε με την έγκριση των πρακτικών. Τις τελευταίες συνεδρίασεις τις τα λάβατε όλοι και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρώ ότι έχουν εγκριθεί και αυτά. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις, οπότε εγκρίνονται. Απόφαση της, ε, των συντονιστών της 22ης ε, Ιουλίου σας έχει αποσταλεί επίσης. Αν έχετε αντιρρήσεις θα πρέπει να τις υποβάλλετε έως σήμερα στις 3 το απόγευμα. Αλλιώς θεωρείτε ότι εγκρίνεται και το πρακτικό της ε, συνεδρίας των συντονιστών. Προχωρούμε λοιπόν στην πρώτη ψηφοφορία για τον ε, προϋπολογισμό για την ε, γνωμοδότηση του Ρόμπερτ Ζήλε. Να δούμε αν έχουν, αν όλοι την ε, κάρτα τους, να κάνουμε μια δοκιμή, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Για να δούμε. Ανοίγει η ψηφοφορία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 Ε, Υπάρχει άλλο πρόβλημα τεχνικό. Να ξανακάνουμε μια δοκιμή. Nein. Gibt es jetzt noch Probleme? Υπάρχουν ακόμη προβλήματα. Όχι, είναι εντάξει. Βγάλτε την λίγο και ξαναπροσπαθήστε. Τώρα εντάξει, ωραία, τέλεια. Και εδώ. Hm? Wer, wer organisiert denn das? Das müssten eigentlich die Universitätsvertreter machen.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 Ωραία. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ψηφοφορία. Τροπολογία 66-24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 66-23. Αποσύρθηκε. 66-25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66-29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ανοίγει η ψηφοφορία. Ποιος δεν έχει την κάρτα του μαζί του. Τώρα λειτουργεί. Εντάξει. Ωραία, άρα λειτουργούν τα πάντα. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουν μία ψήφο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Ωραία, τώρα είναι σωστός ο αριθμός. Λήξη ψηφοφορίας. 34 υπέρ, εγκρίνεται. Nächste ist 6649. 66-49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε κατα... καταπίπτουν 66-50 και 05 και 31 υπέρ. Κατά. Αποχή εγκρίνεται. 66-27 Oral Amendment Υπάρχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις για αυτήν την προφορική τροπολογία. Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Πρέπει να το δούμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 22 κατά, 0 αποχές, εγκρίνεται. 66-51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι υπόλοιποι καταπίπτουν. 66-32 και 66-67. Όχι. 66-52 είναι η επόμενη, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το δούμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Ήταν απαραίτητα να γίνει αυτός ο έλεγχος. 66-53. No, no entiendo por qué que eran compatibles. Δεν καταλαβαίνω σε ποιο βαθμό αυτές είναι συμβατές μεταξύ τους. Εμείς ψηφίσαμε ήδη την 6651 η οποία ήταν συμβατή και γιατί τότε να ψηφίσουμε και την 6632 η, ε, η οποία δεν είναι συμβατή. Διότι εγκρίνεται το 51. Εγκρίθηκε δηλαδή το 6651, γι' αυτό καταπίπτει το 66-06. Bitte mit Mikro. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Eh, Υποτίθεται ότι είναι συμβατές. Είπατε ότι η 036603 καταπίπτει, ενώ η 32 είναι συμβατή με την 51, η οποία ψηφίστηκε και η οποία δεν έχει καταπέσει.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 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6608. Όχι, καταπίπτει. Oral Amendment 6628. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Να κάνουμε ψηφοφορία λοιπόν. Ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6654 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55, υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 66-11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πρέπει να το ελέγξουμε αυτό. Αρχίζει η ψηφοφορία. το ΕΛΚ έχει δύο περισσότερους από ό,τι θα έπρεπε. Συνηθισμένοι είμαστε, αν και νόμιζα ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Ωραία, τώρα ο αριθμός είναι σωστός. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 66-65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 66-13 καταπίπτει. 66-38, όχι καταπίπτει επίσης. 66-02 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66-57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ε, υποψιάζομαι ότι εγκρίνεται, αλλά ξεκινάει η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ έχει έναν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Εντάξει, είναι σωστός πάλι ο αριθμός. Καλώς κάνετε και Προσπαθείτε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 66-43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-01. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66-26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66-03 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και 66-78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Amendments to the draft opinion τροπολογίες στο σχέδιο γνωμοδότησης. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Vote ist geschlossen. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ένα is offen. Το ΕΛΚ έχει πάλι έναν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ακόμη. και εξακολουθεί το ΕΛΚ να έχει έναν περισσότερο. Τώρα είναι εντάξει. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 12 υπέρ. Το 12 ήταν... Ναι, 12. 12 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλαγος. Αρχίζει η ψηφοφορία για το 12. Λήξη geschlossen. Λήξη ψηφοφορίας. Όχι, συγγνώμη. Πάλι το έλκα έχει ένα παραπάνω. Έναρξη ψηφοφορίας. Το προσπαθείτε ξανά και ξανά. Λοιπόν, ξανά. Τροπολογία 12. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Τώρα κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12, 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23. Oral amendment. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική ξεκινά τώρα Το ΕΛΚ έχει πάλι έναν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα είναι σωστός ο αριθμός. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 41 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή Ρόμπερτ Τζίλε. Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Θα κάνουμε λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων με ειδικού για θέματα ασφαλείας της αεροπορίας. και καλωσορίζω τον κύριο Φρανκ Μπρένερ, είναι ε, Γενικός Διευθυντής της Eurocontrol, τον κύριο Σαλβατόρε Σακιτάνο, το προφέρω σωστά, Σακιτάνο λοιπόν, εκτελεστικός γραμματέας της ECIF, της ε, Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας, τον Ζανκόαρλο Μπόνο από την ΙΑΤΑ, περιφερειακό διευθυντή για την ασφάλεια των ε, πτήσεων της ΙΑΤΑ και τον Πάτρικ Κι, εκτελεστικό διευθυντή της EASA, της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να σας ξαναεπισημάνω, ακριβώς επειδή δεν έχουμε αρκετές θέσεις εδώ μέσα ότι έχουμε δημιουργήσει μια αίθουσα δίπλα με οθόνη και με διερμηνία. Να δώσω λοιπόν... Συγγνώμη, παρακαλώ. Ε, voorzitter, goedemorgen. Voorzitter, goedemorgen. Ik zou even van u willen weten hoe precies Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω μία διευκρίνηση. Θα μπορούσατε να μας πείτε ακριβώς αυτό το οποίο θέλετε να κάνουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί θέτω το ερώτημα αυτό. Μερικές φορές κάποιες οργανώσεις κάνουν κάποιες παρουσιάσεις οι οποίες κρατάνε πολλή ώρα. Δείχνουν και πάρα πολλές διαφάνειες και οι παρουσιάσεις αυτές μερικές φορές ε, χρειάζονται για να διαβαστούν πάνω από μία ώρα. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε από τώρα ε, πόσο χρόνο θα δώσετε σε κάθε οργάνωση για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και εμείς τον χρόνο τον οποίο θα αφιερώσουμε στα συγκεκριμένα σημεία και στη γενικότερη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Λόγω ακριβώς του ατυχήματος το οποίο συνέβη στην ε, Μαλαισιανή Αεροπορική Εταιρεία οργανώνουμε την σημερινή ακρόαση. Να σας καθησυχάσω λοιπόν. Ε, κάνουμε το εξής. Τέσσερις ομιλητές έχουμε, δεν θα τους δώσουμε από μία ώρα, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να προγραμματίσουμε τέσσερις ώρες, ενώ έχουμε μόλις τρεις. Έχουμε δώσει περίπου 7 λεπτά στον κάθε ομιλητή. Αφού ολοκληρώσουν τις παρουσιάσεις τους θα κάνουμε μια συζήτηση με τους συντονιστές και στη συνέχεια θα γίνει και ένας κύκλος ερωτήσεων στον οποίο θα μπορέσει να συμμετάσχει ο καθένα. Ωραία, χαίρομαι λοιπόν που το διευκρινίσαμε. Να δώσω λοιπόν πρώτο και κύριε τον λόγο στον κύριο Φρανκ Μπένερ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας κύριε και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι ανάμεσά σας και θα συνεισφέρω όσο πιστεύω καλύτερα στη συζήτησή σας. Το Eurocontrol είναι η ευρωπαϊκή οργάνωση υπεύθυνη για την ασφάλεια των αερομεταφορών και φυσικά θα στηρίξουμε τις προσπάθειές σας. θα σας συστήσω επίσης και τον λεγόμενο μάνατζερ των δικτύων, ο κύριος Τάνερ, ο οποίος ε, κάθεται δίπλα μου. Έχω ορισμένε διαφάνειες εδώ ετοιμάσει που σας εξηγούν ακριβώς τη δομή του ε, ελέγχου του εναρίου χώρου. Το Eurocontrol είναι μια συνδυασμένη οργάνωση πολιτικής στρατιωτικής 40 μελών. Δεν περιλαμβάνουμε μόνο τις 28 χώρες της Ένωσης, αλλά και χώρες πέραν αυτής όπως η Ουκρανία. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι είναι πανευρωπαϊκή οργάνωση το Eurocontrol. Σήμερα θα δούμε ποιος είναι ο ρόλος μας και ο ρόλος κυρίως του διαχειριστή δικτύων. Ε, και στα πλαίσια των ενιαίων ευρωπαϊκών ουρανών του 2004 όπου ζητείται από το Eurocontrol να διασφαλίσουμε την ασφαλή διαχείριση α, ακριβώς ε, των ε, αερομεταφορών. Ο διαχειριστής δικτύων είναι υπεύθυνος για να παρέχει μια συντονισμένη αντιμετώπιση του προγραμματισμού και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των δικτύων. Τα δίκτυα στηρίζουν τους επιχειρησιακούς συμμετέχοντες στα πλαίσια της εκτέλεσης των υποχρεώσεων τις οποίες έχουν αναλάβει και υποστηρίζουν επίσης και τις ε, υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ανάκριση ε, και την έρευνα των αεροπορικών ατυχημάτων. Υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο ε, διαχειρίζεται τη ροή των αερομεταφορών. Το δίκτυο αυτό ε, μπλέκεται επίσης και στον πυρήνα διαχείρισης κρίσεων ε, που δημιουργήθηκε μετά από το, την κατάρριψη του, εμπορικού, ε, του επιβατηγού αεροσκάφους της Παναμέρικαν στη Σκωτία παλαιότερα. Συντονίζει επίσης ε, τις ε, ανταποκρίσεις της κρίσης, είτε είναι η φεστιακή στάχτη αυτό, είτε είναι ένα άλλο τύπου ατύχημα. Βλέπουμε ότι στις δραστηριότητές μας ε, τις υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του πακέτου ενίσχυσης ε, του ρόλου του διαχειριστή του δικτύου. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική και για το μέλλον μας. Θα αναφερθώ τώρα στην διάρθρωση ε, του εναερίου χώρου, πώς οργανώνεται στην Ευρώπη είναι ένας χάρτης που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβαστεί ενιαία, έχει ε, εκατοντάδες μικρές γραμμές οι οποίες δείχνουν τους αεροδιαδρόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια διάρθρωση ανάμεσα στο σημείο αναχώρησης και στο σημείο άφηξης και προσφέρεται στους πελάτες μας που είναι οι αερομεταφορείς. Επιτρέπει στις πτήσεις τους να είναι όσο περισσότερο απευθείας και άμεσες. Έχω εδώ ένα παράδειγμα για ένα πιθανό προγραμματισμό πτήσης από το Λονδίνο στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και ο αερομεταφορέας θα επιλέξει την πλέον κατάλληλη. Ο αερομεταφορέας θα υποβάλει ένα σχέδιο πτήσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως τον αριθμό της πτήσης, τον τύπο του αεροσκάφους, το σημείο αναχώρησης, το σημείο άφηξης, την προτιμόμενη διαδρομή και το ύψος το οποίο προτιμά να πετάψει. Αυτό θα υποβληθεί στον διαχειριστή ε, του δικτύου, θα εξεταστεί ε, για το εάν είναι σύμβατο με ε, κάποιες ρυθμίσεις και θα εξεταστεί αν είναι συμβατό και με τους περιορισμούς μόνιμους ή προσωρινούς. Κάποιοι μόνιμοι περιορισμοί, σαν παράδειγμα, λέγουν ότι ορισμένοι αεροδιάδρομοι χρησιμοποιούνται μόνο για υπερπτήση και όχι για άφηξη και αναχώρηση. Κάποιοι άλλοι προσωρινοί περιορισμοί οφείλονται σε τεχνικές βλάβες των δικτύων ελέγχου των ραντάρ και ε, επίσης προσωρινά ε, κλεισίματα αεροδιαδρόμων κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η μέθοδος ε, βάσει της οποίας επιλέγουν την προτιμόμενη οδό. Εδώ οι συνάδελφοι της ΙΑΤΑ μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να με ε, διαψεύσουν ανάλογα ε, με τους διάφορους παραγόντες που παίζουν ρόλο όπως η κατάσταση του καιρού, οι δυνατότητες μεταφορικές του αεροσκάφους και άλλα θέματα ασφαλείας. Ε, όχι μόνο σε δύο διαστάσεις λοιπόν προγραμματίζει ο αερομεταφορέας αλλά και σε τρεις διαστάσεις. Ε, τα αεριοθούμενα επιβατηγά ε, πετούν συνήθως από 30 μέχρι 45.000 πόδια το, έτσι όπως το ονομάζουμε στα αγγλικά. Αυτό σημαίνει ότι πάνω κάτω στις 4.000 μέτρα. Αυτό, τα τα επίπεδα πτήσης διασφαλίζουν την ασφαλή απόσταση ανάμεσα στα αεροσκάφη. Οι αεροδιάδρομοι μερικές φορές μπορεί όπως είπα να κλείνουν για διάφορους λόγους όπως ε, ο προσωρινός ε, αποκλεισμός του αεροδιαδρόμου λόγω στρατιωτικών εθνικών ασκήσεων Οπότε εκεί ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει αν είναι ασφαλής ο εναέριος χώρος και να τον διαθέσει και στην τρίτη διάσταση, δηλαδή σε επίπεδο ύψους. Εδώ ευθύνε έχουν επίσης ε, και οι συνάδελφοι της ΕΚΑΚ οι οποίοι θα αναφερθούν στο νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει. Τώρα, επανέρχομαι στην τρίτη διάσταση. Μπορεί η αεροδιάδρομη να είναι κλειστή σε χαμηλό επίπεδο, αλλά ανοιχτή σε υψηλό επίπεδο. Μπορεί δηλαδή ε, ο αεροδιάδρομος ο πράσινος να είναι κλειστός, αλλά ο μπλε και ο κίτρινος ανοιχτή. Εάν τώρα ένα αεροδρόμιο ή ένα τμήμα του εναερίου χώρου μιας χώρας κλείσει προσωρινά, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια ανακοίνωση, η λεγόμενη νόταμ. Η διάθεση της συγκεκριμένης πληροφορίας έγκαιρα σε όλες τις χώρες και στους αερομεταφορές. αερομεταφορείς. Οι νόταμ αυτές διανέμονται και είναι διαθέσιμες ε, και για τους ε, Ευρωπαίους χρήστες και για το Eurocontrol που είναι υπεύθυνο για την βάση δεδομένων που συλλέγει όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες σε πραγματικό χρόνο καθίστανται διαθέσιμες στους αερομεταφορείς έτσι ώστε να γνωρίζουν το τι είναι ανοιχτό ή κλειστό κατά τη διάρκεια της πτήσης τους. Ο διαχειριστής λαμβάνει λοιπόν τα νότα αυτά ε, όπως λέει το παράδειγμα εδώ βλέπουμε ότι έχει κλείσει ένας διάδρομος ενός αεροδρομίου και δεν παρέχονται ε, οι υπηρεσίες και έτσι απορρίπτουμε την πρόταση πτήσης εφόσον θέλει να περάσει από εκεί. Λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια και της Task Force του ICAO στην οποία συμμετέχουμε, ε, εξετάζουμε το πώς αυτό το σύστημα, το οποίο είναι αρκετά ασφαλές, θα γίνει ακόμα περισσότερο ασφαλές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και θα πρέπει επίσης ε, οι πληροφορίες τις οποίες θα συλλέξουμε να χρησιμοποιηθούν με τον σωστότερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας κάνω αυτή τη γενική παρουσίαση. Ευχαριστούμε κύριε Μπρένερ για την παρουσίασή σας και περνούμε τώρα στον κύριο Σαλβατόρε Σακιτάνο που είναι ο εκτελεστικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα στα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση με την βοήθεια και του Βέλγου Διευθυντή που είναι το εστιακό σημείο για θέματα ασφάλειας. καθώς τα μεγαλύτερα προβλήματα σχετίζονται με πτήσεις σε ζώνες ε, συγκρούσεων. Η ΕΚΑΚ είναι η πιο παλιά οργάνωση ε, της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκε το 1955. Έχει 44 κράτη-μέλη και ο στόχος είναι να υποστηρίζει την ε, ανάπτυξη ενός ασφαλών και βιώσιμων ενέργειων μεταφορών στην Ευρώπη. Ε, θα επικεντρωθώ, όπως είπε ο κύριος Μπρένον, στο νομικό μέρος και στις ευθύνε των ε, μελών της ε, διάσκεψης για την χρήση του ενέργειου χώρου τους. Αυτά βασίζονται στη Σύμβαση του Σικάγου που υπογράφτηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1944. Δεν θα διαβάσω όλα τα άρθρα. Ήθελα απλώς να τονίσω Ποιε είναι οι κύριε ευθύνε όπως ορίζονται από τη Σύμβαση του Σικάγου. Ε, τα δύο αυτά πρώτα άρθρα, το άρθρο 1 και το άρθρο 9, ορίζουν τις ε, εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση του εναέριου χώρου τους. Ιδίω το πρώτο άρθρο ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος έχει ε, πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον εναέριο χώρο πάνω από το εδάφο, του, πάνω από την επικράτειά του. Το δεύτερο άρθρο, το άρθρο 9, ε, προσδιορίζει την εξουσία ενός κράτους μέλους να περιορίσει ή ε, ε, να απαγορεύσει με ομοιόμορφο τρόπο να υπερίπτεται αεροσκάφη πάνω από την επικράτειά του. Όπως είπε ο κύριος Μπρένερ, τα, το δεύτερο αυτό άρθρο δίνει την εξουσία στα κράτη-μέλη να περιορίσουν την πτήση σε κάποιες ζώνες του ενέργειου τους, όπου υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση με την ασφάλεια των πτήσεων. Μαζί με αυτά τα δύο άρθρα υπάρχει ένα άλλο άρθρο που δεν θα σας διαβάσω, είναι το άρθρο 28, το οποίο ε, δίνει την υποχρέωση στα κράτη-μέλη. Γιατί τα πρώτα δύο άρθρα που σας διάβασα αναφέρονται στις εξουσίες ε, και στα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών πάνω από την επικράτειά τους. Εδώ προβλέπεται μια υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να παρέχουν στην πολιτική αεροπορία υποδομές, υπηρεσίες, ε, ναυσιπλοείας, μετρολογικές υπηρεσίες σύμφωνα με κάποια ε, πρότυπα. Αυτό το άρθρο δηλαδή προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών ε, που αφορούν τον ενέριο χώρο τους. Όπως είπαμε, η οργάνωση του ενέργειου χώρου ε, γίνεται από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη χρήση αυτού του ενάριου χώρου και όλες αυτές οι πληροφορίες ε, παρέχονται ε, στο Aeronautical Information Publication, AIP. Είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους αεροδιοδρόμους, τις αεραχωρήσεις, τις αφήξεις, τις διαδικασίες κλπ. Αλλά όπως είπε ο κύριος Μπρένερ, θα μπορούσαν να ε, εφαρμοστούν κάποιες, κάποιοι προσωρινοί περιορισμοί ανάλογα με τις συνθήκες και οι περιορισμοί αυτοί, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να κοινοποιηθούν μέσω μιας νόταμ, όπως λέμε, notice του airmen. Με βάση λοιπόν αυτά τα πρώτα άρθρα της Σύμβασης του Σικάγο, είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη της ΙΚΑΟ είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια των πτήσεων στον δικό τους ενέργειο χώρο. Πρέπει να παρέχουν πληροφορίες αεροπλοείας και υπηρεσίες σχετικές και πρέπει και μπορούν να περιορίζουν τη χρήση του ενέργειου χώρου τους σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιο ύψος ώστε να εξασφαλίσουν την ε, συνεχή και ασφαλή ε, πτήση. Ε, η αεροπλοεία. Τα ανώταμ, όπως είπαμε, προβλέπονται στο, ε, ή μάλλον οι λεπτομέρειε για τα νότα περιέχονται στο παράδειγμα 15 τη Σύμβασης του Σικάγο, ορίζονται ποιε είναι οι συνθήκε υπό τι οποίε εκδίδονται νόταμ από τα κράτη-μέλη. Το πιο σημαντικό όμω θέμα είναι ποιο είναι υπεύθυνο για την έκδοση μια νόταμ. Μία νότα θα έπρεπε και πρέπει να εκδοθεί από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την χρήση του ενέργειου χώρου, του ενέργειου χώρου του όπως αναφέρουμε προηγουμένως, γιατί μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί λόγω στρατιωτικών ασκήσεων ή άλλων συνδικών που έρχονται σε αντίθεση με την ασφάλεια της αεροπλοείας, αλλά και άλλα συμβαλόμενα κράτη με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες μπορούν να εκδώσουν ε, μια νόταμ που να ενημερώνει τους δικούς του, ε, στους δικούς του μεταφορείς ή μεταφορείς άλλων κρατών μελών για τον ενδυνάμει κίνδυνο σε κάποιες περιοχές και ε, έτσι να τους συστήνει να αποφύγουν την υπέρπτυση σε κάποιες συγκεκριμένε περιοχές. Αυτό προέκυψε μετά από την ε, συντριβή του ε, MH17. Υπάρχει λοιπόν σαφώς ευθύνη του κράτους μέλους για τη διαχείριση του δικού του ενέργειου χώρου. Υπάρχει όμως η δυνατότητα άλλα συμβαλόμενα κράτη με βάση τις διαδέσιμες πληροφορίες να εκδώσουν νόταμ και να ε, ε, ορίζουν ε, περιορισμό συγγνώμη, των πτήσεων σε κάποιες περιοχές του κόσμου. Αν ένα κράτος μέλος που δεν είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση αυτού του συγκεκριμένου ενέργειου χώρου μπορεί να εκδίδει νόταμ για περιορισμό ε, πτήσεις σε αυτή τη συγκεκριμένη ε, χώρα, αυτό πρέπει να βασίζεται σε μυστικές πληροφορίες. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποφεύγεται. Ε, ε, ή δυνατόν. Διότι ε, δεν μπορεί να εκδίδεται μια νότα για κάποιο περιορισμό πτήσεων χωρίς να γνωρίζουν τα άλλα το λόγο. Γι' αυτό μετά τη συντριβή των, το των μελισσιανών αερογραμμών δημιουργήθηκε μια task force για πτήσεις σε εμπόλεμες ζώνες και ο σκοπός είναι να εντοπιστεί ένα σύστημα συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της ε, αεροπορίας η ασφάλεια των πτήσεων πάνω από ζώνες ε, συγκρούσεων. Ο κύριος Μπέρνερ και ο άλλος κύριος είναι μέλη ε, αυτής της Task Force, της ομάδας δράσης και μπορούν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές της. Αυτά βασικά ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες θα θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σακητάνο για την παρουσίασή του και σειρά τώρα έχει ο κύριος Ζανκαλουμόνο από την ε, ΙΑΤΑ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστούμε που προσκαλέσατε την ΙΑΤΑ για να σας παρουσιάσουμε τη δική μας ε, οπτική για, την, ε, για το πώς εκτελούνται και προγραμματίζονται πτήσεις. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ΙΑΤΑ, με Πρόκειται για έναν ε, διεθνή οργανισμό εμπορικό με έδρα το Μόντρεαλ δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε το 1945 και σήμερα αντιπροσωπεύουμε περίπου 135 ε, αερομεταφορείς ε, παγκοσμίω που ανταποκρίνονται, που αντιστοιχούν στο 93% των πτήσεων που πραγματοποιούνται ε, παγκοσμίω. Πρέπει να διασφαλίζουμε διαρκώς την συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία και τους κανονισμούς για να διατηρείται η ε, συμμόρφωση των πιστοποιητικών αυτών θα πρέπει να ε, εφαρμόζουμε όλους τους κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναφερθώ σε όλους τους κανονισμούς, ωστόσο σε ό,τι αφορά την ε, αξιολόγηση του κινδύνου Σύμφωνα λοιπόν με το παράρτημα του ΙΚΑΟ όλοι οι αρμοδιαφορές που έχουν έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, προχωρούν σε αξιολόγηση κινδύνου. Όπως καταλαβαίνετε οι περισσότεροι ε, οι περισσότεροι έχουν ήδη εφαρμόσει αυτή την πρόβλεψη διότι η προθεσμία είναι, ε, εκπνέει σε ένα μήνα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το παράρτημα να μεταφορθεί σε, στο εθνικό δίκαιο των ε, κρατών μελών. Δεν είμαστε οργανισμός, ωστόσο έχουμε πολύ ε, αυστηρούς κανόνες για να δεχτούμε οποιοδήποτε αερομεταφορέα. Και προτού γίνει κάτι τέτοιο, γίνεται ένας επιχειρηματικός έλεγχος για τον έλεγχο ε, της συμμόρφωσης με τις ε, προτινόμενες πρακτικές. Και ένας από αυτούς τους ελέγχους αφορά και τους κινδύνους. Λοιπόν, πρώτου γίνει μέλος κάποιος αερομεταφορέας στην ΙΑΤΑ, ε, διασφαλίζουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν τέτοια συστήματα. Όσον αφορά τους κανονισμούς για την ασφάλεια των ε, πτήσεων, αυτοί ε, βασίζονται στην εθνική νομοθεσία και κάθε αερομεταφορέας είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την εθνική του νομοθεσία. Αυτό που θέλω να τονίσω, που τονίστηκε και από τους συναδέλφους μου πριν, από μένα, είναι ότι κάθε απόφαση για το κλείσιμο ή το άνοιγμα του εναερίου χώρου, καθώς και η υπεύθυνη ε, διανομή ε, των, ε, και έγκαιρη διανομή των πληροφοριών, αφορά τα κράτη-μέλη. Αερομεταφορέας βεβαίως δεν μπορεί να αποφασίσει να κλείσει ή να ανοίξει ένα, ένα αέριο χώρο. Αυτό το κάνουν τα κράτη. Εμείς απλά δρούμε αναλόγως. Πώς γίνεται λοιπόν ο προγραμματισμός των πτήσεων. Όλος ο προγραμματισμός βασίζεται στις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας βεβαίως. Η διαδικασία για τον, για τον προγραμματισμό εγκρίνονται από τις εθνικές αρχές στη βάση όλων των διαθέσιμων επίσημων πληροφοριών όπως είπα μόνιμης, ε, μόνιμου χαρακτήρα, AIP ή προσωρινού χαρακτήρα όπως είναι τα NOTAM, καθώς και όλων των άλλων σχετικών πληροφοριών που ενδέχεται να αφορούν τον εναέριο χώρο μας. Στη συνέχεια προχωρούμε σε αξιολόγηση κινδύνου και αποφασίζουμε αν θα πρέπει να γίνει μια πτήση πάνω, από μια συγκεκριμένη περιοχή ή όχι. Αν ο εναέριος χώρος ε, βεβαίω είναι κλειστός, η απόφαση είναι πολύ απλή, δεν επιτρέπεται η πτήση, οπότε δεν πετούμε εκεί. Αν ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, προχωρούμε σε πτήση σε αυτό την περιοχή μόνο αν ε, από τον αξιολόγηση κινδύνου μας προκύπτει ότι ο κίνδυνος ε, είναι πολύ χαμηλός. Υπάρχει λοιπόν πολύ, ε, μια πολύ, πολύ απλή διαδικασία. Τέσσερα στοιχεία ελέγχει κανείς πριν από την πτήση ως πιλότος. Πρώτον, κοιτούμε την ασφάλεια. Αν δεν είναι ασφαλής μια διαδρομή, τότε δεν ε, πετούμε εκεί. Στη συνέχεια κοιτούμε την, ε, την τακτικότητα. Θέλουμε δηλαδή ε, οι επιβάτες μας να φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους. Στη συνέχεια κοιτούμε τις οικονομικές πτυχές μιας πτήσης, αν δηλαδή συμφέρει, είναι οικονομικά βιώσιμη η πραγματοποίηση μιας πτήσης. Και τέλος κοιτούμε και την άνεση βεβαίως των ε, ε, επιβατών, διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενδεχομένως μια πτήση να είναι ασφαλής, αλλά λόγω αναταράξεων να μην ε, προσφέρει άνεση στους επιβάτες. Να τονίσω εδώ ότι η τελική ευθύνη για κάθε απόφαση που αφορά πτήση στο δικό μας ρυθμιστικό ε, πλαίσιο αφορά τον κυβερνήτη της πτήσης. Όπως είπα, όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, μετά το ατύχημα με, την, ε, με το αεροσκάφος των μαλλισενών ε, αερογραμμών, η ΆΤΑ συμμετέχει, συμμετέχει στην Task Force. Έχουν γίνει δύο συνεδριάσεις μέχρι στιγμής. Περιμένουμε τις επόμενου μήνες να καταλήξουμε σε αποτελέσματα και να καταλήξουμε σε δύο συγκεκριμένα ε, project. Πρώτον, πώς το σύστημα NOTAM που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κοινοποιούνται επίγουσες και κρίσιμη σημασίας ε, πληροφορίες. Δεύτερον, να δημιουργηθεί ένα κεντρικοποιημένο σύστημα για την διανομή τέτοιων ε, πληροφοριών. Βεβαίως, η ποιότητα του συστήματος εξαρτάται πάντοτε και από την ποιότητα των πληροφοριών. Θα συμμετάσχουμε βεβαίως και θα συμβάλλουμε ε, στο μέτρο του δυνατού τις εργασίες αυτής της Task Force σε συνεργασία και με άλλους οργανισμούς, με άλλους ε, υπηρεσίες και με την Flight Safety Foundation. Πρόκειται για μια συνεργασία, σκοπός της οποίας είναι να καταστήσουμε το σύστημά μας ακόμη ασφαλέστερο. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και για τις παρουσιάσεις σας και για το γεγονός ότι ε, σεβαστήκατε το χρόνο και πάμε στον Διευθυντή, τον Πακτρική, τον Διευθυντή της EASA. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Είναι τιμή για μένα το να μπορέσω να κάνω την παρουσίαση αυτή και να πάρω μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Έχω ορισμένες διαφάνειες στα πλαίσια των οποίων θα σας παρουσιάσω την ΕΑΣΑ, ΑΕΣΑ μάλλον, και στον τομέα της ασφάλειας των ε, μέσων αερομεταφορών και των ιδίων των δικτύων αερομεταφορών. Εμείς ε, υιοθετούμε τις γνωμοδοτήσεις μας ε, εν πλήρη ανεξαρτησία από την βιομηχανία ή από τα ευρωπαϊκά όργανα και τα πολιτικά όργανα. Το πιο σημαντικό σημείο σε αυτό το δίκτυο είναι ότι το σύστημά μας αποτελείται από τρεις πυλώνες. Εσάς, ε, την υπηρεσία μας και τα κρατη Όταν εξετάζουμε το πλαίσιο δραστηριοτήτων της ΕΑΣΑ, καλύπτουμε τους διάφορους τομείς των αερομεταφορών. Σε αυτούς τους τομείς ε, έχουμε είτε μια αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως στην πιστοποίηση της ε, αξιοπλόίας είτε μοιρασμένες αρμοδιότητες όπως σαν παράδειγμα στον έλεγχο των αερολιμένων. Ένα παράδειγμα για να σας δείξω το τι κάνουμε στον τομέα των αεροσκαφών, των μέσων μεταφοράς δηλαδή. Εμείς πιστοποιούμε τα αεροσκάφη και τα συστατικά σε εισαγωγικά των αεροσκαφών για όλη την Ευρώπη. Έχουμε έναν μηχανισμό αναγνώρισης των αποτελεσμάτων μας και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και έτσι πιστοποιούμε και τα αεροσκάφη Boeing λαμβάνοντας υπόψη ε, την εργασία της FAA στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και αντίστοιχα η FAA πιστοποιεί ε, τα αεροσκάφη Airbus. Θα ήθελα να πω επίσης ότι πρόκειται για μια αποκλειστική αρμοδιότητα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε οι μοναδικοί στην Ευρώπη που πιστοποιούμε αεροσκάφη. Για να μπορέσουμε εμείς να καλύψουμε τις λειτουργικές ανάγκες που υπάρχουν, έχουμε ένα σύστημα που συλλέγει, αναλύει τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια και σε περίπτωση ε, κατεπήγοντος συμβάντος ε, αμέσως ε, ε, παίρνει αποφάσεις ενημέρωσης ή και αποφάσεις για την ακινησία των συγκεκριμένων τύπων αεροσκαφών. Αυτό είναι κάτι το οποίο συλλέγεται μετά από πληροφορίες των κατασκευαστών, των αερομεταφορέων και των υπηρεσιών των κρατών μελών. Τώρα για την διαχείριση ε, ε, της εναέριας κυκλοφορίας. Εδώ εμείς δεν έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για να πιστοποιούμε σαν παράδειγμα τις υπηρεσίες που ελέγχουν τις, ε, ε, τη, τη, της, τη δράση της πολιτικής αεροπορίας. Εμείς ε, δίδουμε πληροφορίες μέσω των Safety Information Bulletins ε, που ε, τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν είναι υποχρεωτικό να ληφθούν υπόψη από τους συμμετέχοντες στην δραστηριότητα αυτή. Καλύπτουμε μέσω ακριβώς αυτών των Safety Information Bulletin πολλές περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα όπως η Ουκρανία, το Ισραήλ, η Λιβύη, η Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν σχετικά με τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης των εναέριων χώρων των, ε, των εναέριων χώρων των χωρών αυτών. Λοιπόν, μερικές φορές ε, τα κράτη-μέλη δεν δίδουν εύκολα τα στοιχεία τα οποία ζητάμε σαν ΕΑΣΑ. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε μια καλύτερη ροή πληροφόρησης ανάμεσα στο κράτος μέλος και την υπηρεσία μας για θέματα ασφάλειας. Τα πράγματα δεν είναι άσχημα αλλά πρέπει να βελτιωθούν. Απόδειξη αυτού είναι ότι για όλα τα bulletin τα οποία έχουμε δημοσιεύσει μέχρι τώρα για το Ιράκ, Αφγανιστάν, Ισραήλ κτλ. Οι πληροφορίες έρχονται αποκλειστικά από την Αμερικανική κυβέρνηση λόγω της συμφωνίας που έχουμε αμοιβαία συνδρομής στα θέματα ασφάλειας. Λοιπόν, το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε συμβατοί με τις δραστηριότητες του ΙΚΑΟ παγκόσμια. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, έκφραση συγκεκριμένης ανάγκης ενός συστήματος προειδοποίησης στην Ευρώπη που να καλύπτει όλους τους κλάδους. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να ε, συγκεντρώνεται κυρίως στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών γιατί εδώ ακριβώς ε, υπάρχει θέμα και επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές αρμοδιότητες των διαφόρων τμήματων, να υπάρχει σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων. Οι πληροφορίες θα πρέπει να υπακούν σε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για να γίνει αυτό απαιτείται η σωστή εμπλοκή ε, των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών και φυσικά και η συμμετοχή του Eurocontrol στα πλαίσια της συλλογής και στη συνέχεια διάδοσης των πληροφοριών αυτών. Εμείς πιστεύουμε σαν υπεύθυνοι για θέματα ασφαλείας ότι μπορούμε να παίξουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο ε, για την δημιουργία αυτού του συστήματος προειδοποίησης. Έχουμε τα μέσα τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουμε να ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκομένους και τα μέσα άμεσης ε, χρήσης ε, έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή εξέλιξη στο μέλλον. Θα θέλαμε λοιπόν να σας προτείνουμε να μας βοηθήσετε εσάς και τα ευρωπαϊκά όργανα. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται βέβαια ε, με σωστό συντονισμό με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε για να υπάρξει ένα σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να πετύχουμε αρκετά πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες, η βιομηχανία, οι επιβάτες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να είναι βέβαιοι ότι η δραστηριότητα αυτή είναι μια ασφαλής δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Πριν δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστές, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Μάθιου Μπόλτουεν είναι ο αρμόδιος ε, διευθυντής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην πρώτη συνεδρίαση της ε, εντελώ καινούργια αυτής ε, Επιτροπής Μεταφορών. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο για τον ρόλο του και σας συγχαίρω επίσης που διαλέξατε ένα τόσο σημαντικό θέμα για την πρώτη συζήτηση για τις ε, εναέριες μεταφορές. Βέβαια αυτό σχετίζεται με το τραγικό ατύχημα του MH17. Θα ήθελα να πω εντό παρενθέσεως ότι ήταν πολύ δύσκολο το καλοκαίρι όσον αφορά την πολιτική αεροπορία. Ε, χάσαμε τα δύο MH17, όπως ξέρουν πολλοί συνάδελφοι εδώ. Άλλο ένα τρομερό ατύχημα, H504 ε, στο Μαλί. Είχαμε το έμπολα που είχε επιπτώσεις και για την ε, πολιτική αεροπορία και ακόμα ένα ε, Ισλανδικό ηφαίστειο ε, που προς το παρόν παραμένει ήρεμο. Δεν θέλω να επαναλάβω κανένα από τα σημεία των εξαιρετικών παρουσιάσεων που ακούσαμε γιατί θα ήταν σημαντικό να περάσουμε γρήγορα στις ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω πολύ σύντομα κάποια από τα σημεία που ακούσαμε ήδη. Το πρώτο βασικό σημείο που ακούσαμε είναι ότι οι αποφάσεις για την ασφάλεια των αέριων παραμένει ευθύνη των κρατών. Αυτό είναι κανόνας του ΙΚΑΟ. Το είπε πολύ ε, καθαρά ο Σαλβατόρε που μας ε, το συσχέτισε με τη σύμβαση του Σικάγο και αυτός είναι ο πυλώνας γύρω από τον οποίο λειτουργούμε. Το δεύτερο σημείο, για είμαστε πολύ ξεκάθαροι, είναι το εξή ότι στην πραγματικότητα τα κράτη-μέλη μπορεί στην πράξη να μην είναι σε θέση να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό και, πολύ, και οι πολύ επίγουσες συζητήσεις που έγιναν τον Αύγουστο στο ΙΚΑΟ για να αναθεωρηθούν οι κανόνες αυτοί και να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Βεβαίω, θα πρέπει επίση να καταλάβουμε ότι ο κίνδυνο είναι ότι η, η εκτέλεση αυτή τη υποχρέωση είναι πιο δύναμη κατά πάσα πιθανότητα σε περιοχέ και σε κράτη όπου είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν οι, κίνδυνοι. Είναι ε, πολύ λιγότερο πιθανό να έχουμε στις περιοχές αυτές η ικανοποιητική ε, αξιολόγηση του κινδύνου. Και δεν μιλάω για την ειδική περίπτωση της Ουκρανίας εδώ πέρα, μιλάω για τον συστήμα συστημικό κίνδυνο που γίνεται πολύ πιο σαφής. Τρίτο σημείο. Ε, ακούσατε τις απόψεις των αερομεταφορεών από την ΙΑΤΑ και τις ε, πολύ αυστηρές υποχρεώσεις που επιβάλλουν ε, στα μέλη τους οι ίδιοι για την αξιολόγηση του κινδύνου. Είναι σαφές όταν είναι κλειστός ο αέριος χώρος δεν υπάρχει πτήση, όπως είπε ο κύριος. Πτήση μόνο όταν ο κίνδυνος είναι αποδεκτός, το επίπεδο του κίνδυνου είναι αποδεκτό. Αλλά και πάλι το ερώτημα είναι οι αερομεταφορείς έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να το κρίνουν. Και εδώ πάλι έχουμε ένα ε, φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πάτρικ Κι της ΕΑΣΑ έκανε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Και συμφωνούμε ότι ενώ τα κράτη έχουν αυτές τις υποχρεώσεις, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και προς την ε, ΕΑΣΑ και προς τον διαχειριστή ε, της ασφάλειας των αερομεταφορών. Και αυτό είναι το ε, κυριότερο σημείο. Η συλλογή και η διάχυση των πληροφοριών. Αλλά και η ΕΑΣΑ και ο ε, φορέας που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των πτήσεων ε, είναι υπεύθυνοι για την ε, διάδοση αυτών των πληροφοριών με τα μπουλέτιν που ακούσαμε. Τώρα, για να έρθω σε ένα άλλο σημείο που ανέφερε ο Πάτρη, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων ε, επιβατών. Πρέπει να συνδυάσουμε γνώσεις και ε, μυστικές πληροφορίες. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε κυρία Πρόεδρε, δεν έχουμε στρατιωτικό σκέλος, δεν έχουμε στρατιωτικές ε, υπηρεσίες πληροφοριών στις οποίες να μπορούμε να βασιστούμε. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες είναι πολύ σημαντική. Αυτό θα συμπληρώσει την ενημέρωση που έχουμε και ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Eurocontrol και για τους αερομεταφορείς. Και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, είτε ε, σαν βάση είτε για προαιρετική είτε για υποχρεωτική ε, αποφυγή κάποιων ε, πτήσεων. Ξέρω ότι οι αερομεταφορείς μπορούν να απαγορεύσουν την πτήση σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Μπορεί να υπάρχει εθνική απαγορεύση όταν υπάρχει co-sharing κλπ. Κάτι άλλο που προέκυψε στην ΕΚΑΟ και θα ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο πιστεύω ε, έχει να κάνει με τη διαφάνεια προς τους ε, επιβάτες. Καταλαβαίνω ότι είναι ε, ελκυστικό αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να σας προειδοποιήσω το να ενημερώσουμε εκ των προτέρων τους επιβάτες για ποιον αεροδιάδρομο θα χρησιμοποιήσουν, πάνω από ποιες περιοχές συγκρούσεων θα πετάξουν κλπ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να οργανωθεί. Και καταλαβαίνω το αίσθημα των ε, αερομεταφορέων. Ε, όταν αγοράζει κανείς το εισιτήριο θα πρέπει να ξέρει το σχέδιο πτήσης. Τα σχέδια πτήσεων ε, μπορεί να αλλάξουν Να πάσα στιγμή για πολύ βάσιμους επιχειρησιακούς λόγους. Ή ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να δημοσιεύουν ε, τι πληροφορίε αυτέ. Με αυτό δεν θα αυξήσει τον κίνδυνο και την ευαλωτότητα ε, τη πτήση. Δεν θα γίνει πιο εύκολο στόχος. Και όλα αυτά τα θέματα που είναι αρκετά ε, περίπλοκα, ε, ήθελα απλώ να επισημάνω κάποιους από τους κινδύνους. Ε, ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και προχωρούμε τώρα στο γύρο των συντονιστών. Τέσσερα λεπτά έχει στη διάθεσή του ο κάθε συντονιστής και στη συνέχεια, ανάλογα με το πόσο μιλητές θα έχουμε, θα δώσουμε δύο έως τρία λεπτά. Για το ΕΛΚ λοιπόν ο εκπρόσωπος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε τη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους εμπειρογνώμονες για τις παρουσιάσεις τους. Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω, ένα πρώτο σχόλιο. Μας μιλήσατε για το τι ισχύει σήμερα, τι υπάρχει σήμερα, τι διαδικασίες υπάρχουν, τι ευθύνες, ε, κατανομή ευθυνών υπάρχει, αλλά δεν έχουμε πει ακόμα το τι ε, πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα μετά από το ατύχημα του μηνός Ιουλίου είναι ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το οποίο θίγει την ασφάλεια των πτήσεων η οποία είναι η πρώτη ανησυχία, η βασική προτεραιότητα όλων των αερομεταφορών γενικότερα. Νομίζω λοιπόν ότι στην παρούσα φάση δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας στη συγκεκριμένη πτήση και δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτής της παράληψης ήταν τραγικά αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ένα επίσης τραγικό παράδειγμα, ότι απαιτείται να υπάρξει καλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτή τη φάση των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Δυστυχώς όμως τα κράτη-μέλη είναι πάντα εναντίον αυτού του συστήματος, ε, του συστήματος ε, που λέγεται Single European Sky. Έχω λοιπόν μία πάρα πολύ απλή παρατήρηση να κάνω. Γνωρίζουμε όλοι το τι ακριβώς συνέβη στην Ουκρανία. αλλά ακόμα και μετά από το τραγικό αυτό συμβάν δεν υπήρξε μία συνεκτική ανταπόκριση των ευρωπαϊκών οργάνων. Υπήρξαν πολλές πληροφορίες από πλευράς των Ουκρανών, από πλευράς των Ρώσων, ε, κάτι το οποίο οδήγησε και σε συγκρούσεις μεταξύ τους σε επίπεδο ενημέρωσης γιατί τα στοιχεία ενημέρωσης που παρουσίασαν ήταν αντιφατικά. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης τίποτα. Έχω λοιπόν ένα πολύ απλό ερώτημα να σας θέσω. Τι θα κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε ε, να ληφθούν μέτρα, νομοθετικές ρυθμίσεις, διαδικασίες ε, στο μέλλον για να εμποδιστεί η επανάληψη αυτών των απαράδεκτων καταστάσεων. Έχει μεγάλη σημασία ο επιβάτης να αισθάνεται ασφάλεια, να γνωρίζει ότι είναι ασφαλής. Είτε ε, η περίπτωση της Ευρώπης είτε της Ασίας πρέπει αυτό να μπορεί να το κάνει με συνθήκες ασφαλείας. Πώς λοιπόν θα αντιδράσετε και πώς θα αντιδράσετε γρήγορα γιατί το να λέμε ότι τα κράτη-μέλη φταίνε Ε, το κράτος μέλος, αν και δεν ήταν κράτος μέλος στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν ένα κράτος μέλος μόνο του αεροκοντρόλ. δεν σεβάστηκε ίσως τις διαδικασίες και τα λοιπά. Ε, δεν αρκεί να λέμε ότι εμείς απλά προειδοποιήσαμε ότι στην περιοχή αυτή ε, έχει μια σύγκρουση. Δεν φτάνει αυτό, δεν είναι επαρκές ε, για την ασφάλεια των επιβατών. Οφείλετε λοιπόν να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις και απευθύνομαι εδώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις ευθύνες τους σε σχέση με τη συλλογή των πληροφοριών, την αξιολόγησή τους και τη λήψη των ξεκάθαρων αποφάσεων. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να υπερίπταται μια ζώνης ε, ανοιχτής σύγκρουσης. Ο κύριος Μπρένεν μας παρουσίασε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για να αποφεύγει κανείς ε, ε, ε, μια τέτοια περιοχή. Η αλλαγή ύψους δεν αρκεί. Ποιες είναι οι προτάσεις που θα κάνετε στο μέλλον λοιπόν για να αποφευθεί επανάληψη αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Ο έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχικά να πω βεβαίως ότι αυτό που συνέβη τον Ιούλιο ήταν μια καταστροφή Εκφράζουμε λοιπόν και εμείς ε, τα συλληπιτήριά μας σε όσους έχασαν συγγενείς και φίλους. Έχω πολλά ερωτήματα, πέντε συγκεκριμένα. Ξεκινώ με ένα και μπορεί να το απαντήσει όποιος θέλει ή όποιος μπορεί. Μετά το δυστύχημα αυτό δημιουργήθηκε μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων που ε, τον Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει τα πορίσματά της και θέλω να ρωτήσω σε σχέση με αυτό σε ποιο βαθμό έχετε συνεργαστεί με αυτή τη διεθνή ομάδα. Δεύτερο ερώτημα προς την Eurocontrol, τον κύριο Μπρένερ και τον εκπρόσωπο της ΕΑΣΑ. Αρχές ε, Ιουλίου φέτος υπήρξαν διαταραχές ε, στον ενεάριο χώρο πάνω από τις Άλπεις εξαιτίας μιας πηγής βλάβης και αυτό κατέστησε αδύνατη την ε, πραγματοποίηση πτήσεων. Μήπως ε, αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε αόρατη η πτήση MH17. Η Austria Control δεν ενημερώθηκε για το θέμα αυτό και έχω και ένα ερώτημα για τη Eurocontrol. Από αρχές Ιουλίου, αν έμαθα σωστά, ο ενέωριος χώρος πάνω από την Ανατολική Ουκρανία ήταν κλειστός, ωστόσο το κλείσιμο αυτό αφορούσε τα 32.000 πόδια και η πτήση αυτή πετούσε στα 33.000 πόδια. Είναι ορθό αυτό και αν ναι, ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζουμε από το γεγονός αυτό. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Φοντάλ έχει το λόγο για το ECR. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> πρόεδρε, είναι τα γενέθλιά μου σήμερα πρέπει να σας πω και χαίρομαι πάρα πολύ που εγώ είμαι σε θέση να τα γιορτάσω. Υπάρχουν όμως οι 300 τόσοι επιβάτες του MH17 που ποτέ πια δεν θα ε, ξαναγιορτάσουν τα γενέθλιά του, γιατί κάποιοι τρελοί που είχαν ε, πυράβλους στη διάθεσή τους έριξαν ε, στην τύχη ε, χωρίς να ε, σκέφτονται ότι υπάρχει και η πολιτική αεροπορία. Ε, 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 96 ήταν ε, Ολλανδικής υπηκότητας. Ε, ε, σχεδόν, ε, ή 196 μάλλον. Ο καθένας σχεδόν στη χώρα μου ξέρει κάποιον που ήταν σε αυτή την πτήση. Είναι μια εθνική τραγωδία για μας και δεν είναι καν ε, δυνατόν να εντοπιστούν οι σωροί των θυμάτων. Τα σώματά τους παραμένουν εκεί στον τόπο της συντριβής. Ε, και δεν είναι ε, δυνατόν ε, καν να γίνει συστηματική διερεύνηση του ατυχήματος αυτού γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στον τόπο της συντριβή. Αυτό ήταν μια καταστροφή φυσικά για όλους τους επιβάτες της τήσης αυτής, για όλες τις χώρες που έχασαν τους υπηκόστους και μια καταστροφή για την πολιτική αεροπορία. Την περασμένη εβδομάδα συζητήθηκε το θέμα αυτό και πληροφορηθήκαμε ότι στις, ότι στη... την... Ε, μέχρι τις 17 Ιουλίου, 14, 15 και 16 και 17 Ιουλίου είχε υποβάλει το σχέδιο πτήσης αυτό η αεροπορική εταιρεία στην Eurocontrol και στις 17 Ιουλίου ε, εγκρίθηκε αυτό το σχέδιο πτήσης, ακριβώς το ίδιο σχέδιο πτήσης. Και η μόνη διαφορά υποτίθεται ότι ε, θα ήταν ότι θα περνούσαν από τον αεροδιάδρομο 350 στον αεροδιάδρομο 330. Ενέκρινε λοιπόν αυτό το σχέδιο πτήσης Eurocontrol. Ε, στις 14 Ιουλίου οι British Airways είχαν ήδη αποφασίσει να μην ε, πετάνε πάνω από αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι ακριβές. Είχαν ε, αποφασίσει όντως οι British Airways από τις 14 Ιουλίου να μην πετάνε πάνω από αυτή την περιοχή. Και γιατί δεν είχε κοινοποιηθεί η πληροφορία αυτή στις άλλες ε, αεροπορικές εταιρείες. Και ποιο είναι το σχέδιο που έχει Eurocontrol για την βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων. Γιατί... Ε, δεν ενημερώθηκαν όλες οι άλλες εταιρείες. Γιατί δεν ήρθε σε επαφή η Eurocontrol με την British Airways για να ρωτήσει ποιος ήταν ο λόγος που άλλαξαν ε, τα δρομολογιά τους. Ε, ποιος ήταν ο λόγος. Ε, υπάρχουν ε, προφανώς τεράστια κενά στο όλο σύστημα. Ε, τεράστια κενά στον τρόπο που ε, διατίθενται ε, οι πληροφορίες. Κάποια κράτη έχουν καλύτερες πληροφορίες από άλλα. Υπάρχει λοιπόν ε, μια ένα, τεράστια, ένα τεράστιο κενό εδώ. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρέπει οι πληροφορίες να κοινοποιούνται με το σωστό και έγκαιρο τρόπο. Όπως είπα, οι άνθρωποι που είχαν την ατυχία να βρίσκονται σε αυτή την πτήση ε, δεν θα ξαναγιορτάσουν ποτέ τα γενέθλιά τους και το ίδιο και οι οικογένειές τους. Κάποιοι πρέπει να μοιραστούν και να αναλάβουν αυτές τις ευθύνες. Ευχαριστώ ακόμη και αν η συσχέτιση που κάνατε με τα γενέθλιά σας είναι αρνητική, ε, παρόλα αυτά θέλω να σας ευχηθώ. Ελπίζω να μπορώ να το πω αυτό και εκ μέρους όλης της Επιτροπής. Ε, Άλντε, και Ζήνε να έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ένα πρακτικό ερώτημα. Ως μέλη της ε, Επιτροπής μπορούμε να, μπορούμε να λάβουμε αυτές τις παρουσιάσεις που παρακολουθήσαμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ, απλά ήθελα να το πω. Μια γενική παρατήρηση και Μπρένερ, είπατε ότι ο προγραμματισμός της πτήσης γίνεται με όσο πιο άμεσο τρόπο γίνεται. Δεν μπορώ ωστόσο να αποφύγω να σας πω ότι ο ευρωπαϊκός, ε, ευρωπαϊκός ουρανός αν τον είχαμε, θα μπορούσε να διασφαλίσει να γίνονται ακόμα πιο άμεσες πτήσεις και ακόμα περισσότερος συντονισμός, ιδιαίτερα όσον αφορά και τη διασφάλιση την, ε, της ασφάλειας των πτήσεων στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολλές οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις που πρέπει να συντονιστούν. Και το άλλο μου ερώτημα μου είναι το εξής. Βεβαίως όλοι ε, έχουμε στο νου μας αυτήν την πτήση, την MH17. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποιος είναι ο υπεύθυνος τελικά για το γεγονός αυτό, διότι θα ε, εξεταστεί σίγουρα και ποιος θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί ε, υπεύθυνοι. Υπεύθυνο είναι και ο κυβερνήτη. Εκείνο όμω φέρει την ευθύνη για όσα γνωρίζει, άρα θα πρέπει να έχει ενημερωθεί. Σημαίνει αυτό ότι και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα, διότι πρέπει να περιορίζουν τι πτήσει σε ορισμένε περιοχέ η Ουκρανία. Δεν το έκανε. Άρα ποιο είναι υπεύθυνο, είναι ο κυβερνήτη υπεύθυνο, είναι η Ουκρανία υπεύθυνη, διότι δεν είχε εκδώσει απαγόρευση πτήσεων για τη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Πούτιν, και αυτό μπορεί να πει κανεί ε, ότι είναι υπεύθυνο. Η EASA είναι υπεύθυνη βεβαίω για την Ευρώπη, για την ασφάλεια του εναέριου χώρου στην Ευρώπη. Αυτό είναι γενικά σωστό. Αλλά μήπως τελικά έχουμε πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι δεν συντονίζονται επαρκώς στην Ευρώπη. Το ξέρω ότι έχετε πολύ καλές υποδομές, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά όργανα, πάρα πολλοί οργανισμοί, υπηρεσίες που ασχολούνται με την ασφαλεία των πτήσεων και ο κυβερνήτης θα πρέπει να είναι δικτυωμένος με όλους αυτούς. Άρα το ερώτημα μου είναι μήπως τελικά έχουμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και οργανισμών. Και το τελικό μου ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να αποτρέψει τρομοκρατικές ενέργειες ή πώς μπορεί κανείς να προβλέψει τέτοιου είδους ενέργειες ή υπάρχουν και ενέργειες τις οποίες δεν μπορεί κανείς να τις επηρεάσει με κανέναν τρόπο. Και γι' αυτό και το ερώτημά μου είναι ε, η Task Force της ICAO γιατί δημιουργήθηκε τώρα. Υπήρχε και στο παρελθόν κάτι ανάλογο. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι υπήρχε μια τέτοια task force. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μόλις τώρα δημιουργήθηκε μια τέτοια ομάδα. Και το τελικό μου ερώτημα. Εμείς πώς έχουμε πρόσβαση, έχουμε πρόσβαση ε, στις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών όσον αφορά τους κινδύνους που ε, ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν ίσως και αλληλεπιδράσεις που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε προκειμένου να ενισχύσουμε την ασφάλεια των πτήσεων. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος για την Kiitoksia puheenjohtaja, ευχαριστώ συνάδελφε. Όλα τα ατυχήματα φυσικά είναι κάτι το οποίο προκαλούν, προκαλεί λύπη. Φυσικά θα μπορούσε κανείς να, ε, να ονειρευτεί ότι μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω και να διορθώσει ε, τα πράγματα αναδρομικά, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Με τις πληροφορίες τις οποίες πήραμε μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να πούμε στους επιβάτες πλέον και ιδιαίτερα στους συγγενείς των θυμάτων, ότι ζούμε σε έναν κόσμο που διασφαλίζεται πλήρως ε, η αερομεταφορά επιβατών. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξαναγίνει αυτό το οποίο συνέβη. Πολύ συγκεκριμένα. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε ανεξαρτήτως των προβλημάτων που υπάρχουν στον κόσμο οι επιβάτες ε, θα είναι ε, σίγουροι ότι ε, όταν ξεκινούν το ταξίδι τους ε, θα φτάνουν και στον προορισμό τους. Χρειάζονται περισσότερα μέτρα και πιο συγκεκριμένα μέτρα. θα πρέπει ε, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των αερομεταφορών διαφορετικά από ό,τι μέχρι σήμερα. Κανένας δεν είναι σε θέση να πει ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα συστήματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ίσως σήμερα να υπάρχουν και πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι οι οποίοι κατανέμουν τις αρμοδιότητες χωρίς τελικά να υπάρχει ένας τελικός υπεύθυνο. Οι επιβάτες θέλουν ένα δικαίωμα να τους διασφαλίσουμε, το δικαίωμα του να ταξιδέψουν με ασφάλεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή μας μάλλον, που οργάνωσε τη συγκεκριμένη ακρόαση. Γιατί σήμερα στόχος μας είναι να φροντίσουμε ε, για να μην επαναληφθεί η καταστροφή ε, της πτήσης των Μαλαισιανών αερογραμμών. Έχω αρκετές ερωτήσεις ε, ε, να κάνω γιατί σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή νομίζω. Η πρώτη ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν με τέτοια συμβάντα τα οποία αυτή τη στιγμή διεξάγονται στην Ουκρανία ε, πώς στάθηκε αδύνατο να εκτιμήσουμε σωστά την επικίνδυνοτητα του εναερίου χώρου. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το γιατί η Ουκρανία και η Ρωσία δεν έστειλαν όταν Και αν έστειλαν όταν τότε τι είδους πληροφορίες περιλάμβανε. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι εδώ και αυτό το είπαν. Υπάρχουν η πολιτική αεροπορία, τα κράτη-μέλη, η ΑΕΣΑ. Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι ε, έπαιξαν το ρόλο τους, ήταν αρκετά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί ή μήπως θα πρέπει να πούμε ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία έχουν κατά κάποιο τρόπο τελικά την ευθύνη αξιολόγησης του επίπεδου του κινδύνου. Τίθεται λοιπόν το θέμα της ευθύνης. Είναι ένα σοβαρό θέμα το ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος. Το θέμα είναι το θέμα εδώ των κυρώσεων το οποίο τίθεται βέβαια. Πώς θα αξιολογήσουμε τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν για να μην ξανασυμβεί αυτό το οποίο συνέβη. Εσείς λοιπόν μπορείτε να μας πείτε τι έχετε στο νου σας, ε, τι ε, τομείς, τι παιδεία ανοιχνεύεται έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί η καταστροφή που συνέβη. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά θα ήθελα να μάθω το πώς θα ενισχύσετε την συγκέντρωση και το συντονισμό, τη συγκέντρωση των στοιχείων και τον συντονισμό τους. Πώς θα το πετύχετε αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα σύμβαση, συνθήκη με τα κράτη-μέλη. Ο εκπρόσωπος της ΕΑΚ είπε προηγουμένως ότι υπάρχουν 44 μέλη. Ε, θα μπορούσατε να δώσετε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει ε, μεγαλύτερο ρόλο ή μια εξωτερική υπηρεσία για τον συντονισμό. Δεν είναι προτάσεις αυτό που κάνω τώρα, είναι ερωτήσεις. Αλλά διαρωτώ με αν έχετε σκεφτεί αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Το να ενισχύσει κανείς ε, την αποστολή της ΕΑΣΑ, της ΑΕΖΑ, ε, είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο να γίνει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι. Αλλά παρόλα αυτά ε, ποιοι είναι οι τομείς τους οποίους εσείς εξετάζετε ε, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ Λούντγκρεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ οι μαλλισσινές αερογραμμές, η πτήση των μαλλισσιών ε, αερογραμμών στην αίρια του Ντονέτσκ ε, τον Ιούλιο περιβάλλεται από αντικρώμενες πληροφορίες διότι ακούστηκε πολλές πλευρές ότι ε, το, το, η κατάρρευση έγινε με πυράβλους Μπουκ των φιλορώσων αυτονομιστών υπήρξαν και πληροφορίες ότι υπήρξε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος κοντά στην, ε, στο αεροσκάφος MH17. Έκτοτε δεν γνωρίζουμε τίποτα ούτε για το μαύρο κουτί ούτε τίποτα και χρειάζεται, περνά πάρα πολύ χρόνος σε σύγκριση ιδιαίτερα και με άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Οπότε πρέπει να είμαστε σαφείς προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων επιβατών. Αλλά πώς μπορούμε να αποκτήσουμε τις πληροφορίες, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την κατάσταση των ε, ερευνών που γίνονται. Το γραφείο της Ουκρανίας ζήτησε από την EASA να ορίσει υπεύθυνο να ε, συμμετάσχει στην ε, ομάδα που συνεδρίασε στις 21 Ιουλίου. Η το EASA θα συνεχίσει βεβαίως να ε, συμβάλλει στις εργασίες του Ολλανδικού Γραφείου. Βεβαίως συμμετέχουν μια σειρά από χώρες, Μαλαισία, Αυστραλία, ε, Ουκρανία, αλλά μάθαμε ότι το, η e δεν είχε λάβει πληροφορίες για τον περιορισμό που είχαν εκδώσει οι Ουκρανικές αρχές. Δεύτερο ερώτημα. Αυτού του είδους οι πληροφορίες Τι γίνεται με τους, με αερομεταφορείς, ε, λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις, οι αρχές εγκρίνουν αεροδιαδρόμους ανεξάρτητα από την ή λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που ισχύει ε, σε διάφορες χώρες. Η, η ΆΣΑ ε, έχει αρμοδιότητα ε, για τα αεροσκάφη από την Ευρώπη. Τι συμβαίνει όμως με ε, τις ε, αεροπορικές εταιρείες άλλων χωρών. Τι συμβαίνει με την ασφάλεια των επιβατών. Ακούμε ότι η Άσα διανέμει συστάσεις και πληροφορίες ασφάλειας μέσω των AIP. Τέταρτο ερώτημα. Τι συμβαίνει με τους επιβάτες. Πώς θα ενημερώνονται εκείνοι σχετικά με την ασφάλεια της διαδρομής που θα ακολουθήσουν. Οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για την EASA. Και τι συμβαίνει με τον πραγματικό έλεγχο της ασφάλειας των επιβατών είναι απαραίτητη η Άσα τελικά ή μήπως θα ήταν καλύτερο τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται την ασφάλεια του εναέριου χώρου τους χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετα κόστη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Προτού δώσω το λόγο στους υπόλοιπους, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στους ε, ομιλητές μας σήμερα να απαντήσουν στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ξεκινάμε με την ίδια σειρά. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές και τις παρεμβάσεις. Για το θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, και θα ξεκινήσω με αυτό, και τις περαιτέρω εξελίξεις, είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε στο θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, βελτιστοποιώντας στην Ευρώπη το σχεδιασμό των ε, διαδρομών, των δρομολογίων. Ε, έχουμε σχέδια βελτιστοποίησης, έχουμε μειώσει το μήκος των διαφόρων διαδρομών, αλλά θα είναι ε, σημαντικό να προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα, όπως προτείνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι περιμένω να δω μεγαλύτερη υποστήριξη από το Κοινοβούλιο σε αυτήν την ε, πορεία δράσης, για καλύτερη βελτιστοποίηση και λιγότερο κατακαιρματισμό. Τώρα, στην ερώτηση γιατί η ε, Eurocontrol δέχτηκε αυτό το σχέδιο πτήση. Η ε, Eurocontrol ελέγχει όλα τα σχέδια πτήση που εκδίνονται στην Ευρώπη, από προς μέσα στην Ευρώπη, σύμφωνα με, ε, τα δημοσιευμένα που υπάρχουν. Όπως είπε ο Σαλβατόρε, αυτό βασίζεται στις εκδόσεις Νόταμ. Η λοιπόν των μαλαισιανών γραμμών σχεδίαζε να ακολουθήσει μία διαδρομή και σε ένα ύψος που ήταν ανοιχτό στις πτήσεις. Και δεν υπήρχε κανένας περιορισμός σε αυτό το ύψος πτήσης. Κάτω από αυτό το ύψος είχαν κλείσει ε, οι αεροδιάδρομοι από την Ουκρανία. Αλλά ε, το σχέδιο πτήσης ήταν πάνω από, την, ε, από το ύψος όπου υπήρχε η απαγόρευση πτήσης οι πληροφορίες αυτές ήταν διαφανείς, ήταν διαθέσιμες για όλους. Το πρόβλημα ήταν ότι τέτοιου είδους κλεισίματα ή περιορισμοί έχουν κάποιο υπόβαθρο. Κάποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ένα κράτος μέλος για να καταλήξει στην απόφαση ε, για το κατά πόσο μια περιοχή του ενέργειου χώρου θα πρέπει να είναι ε, ανοιχτή ή όχι. Και σε αυτό αναφέρθηκε και ο Πάτρικ Κι ότι αυτές οι πληροφορίες ε, υπάρχουν σε ε, μεμονωμένη βάση, είτε, σε, ε, είτε βάση διμερών, συμφωνιών ή σε μεμονωμένη βάση. Δεν είναι κοινέ γνώσεις και πληροφορίες αυτές. Άρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε Ποιος ήταν ο συλλογισμός εκείνη την εποχή των Ουκρανικών αρχών, γιατί έκλεισαν τον ενάριο χώρο κάτω από αυτό το ύψος και όχι πάνω από αυτό το ύψος. Και ε, αυτές είναι οι πληροφορίες που οδήγησαν σε αυτή την αξιολόγηση του κινδύνου. Ε, αν τις είχαν αυτές τις πληροφορίες, ε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό η ΚΑΟ θα πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα ως προς το θέμα αυτό της ε, ε συλλογής πληροφοριών. Τώρα για το θέμα της ε, των πληροφοριών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να, που, που έχουν αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τις χρησιμοποιούν για τη διαχείριση κινδύνου και εμείς ως διαχειριστές θα, πρέπει, ε, θα, θέλαμε να έχουμε και εμείς αυτές τις πληροφορίες για να ε, ελέγχουμε τη συνέπεια των αποφάσεων. Ε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια ατυχήματα αν δεν μπορούμε να βασιστούμε στις, ε, στα διδάγματα από την τραγωδία ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Η κοινοποίηση, το μοίρασμα αυτών των πληροφοριών είναι ε, πολύ σημαντική. Ε, είπαμε ότι δεν παίρνουμε στρατιωτικές φύσης πληροφορίες, παρά μόνο σε αποσπασματική βάση. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια σημαντική βελτίωση. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και ε, στρατιωτικές πληροφορίες. Ε, το να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη σε κάποιο βαθμό να διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες ε, είναι ένα βήμα το οποίο συζητάμε στην Task Force. Ο κύριος Σαλβατόρος Σακητάνου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η πολιτική αεροπορία εξορισμού είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Είναι μια δραστηριότητα που δεν περιορίζεται σε μια περιοχή ή σε ένα κράτος, αλλά είναι μια διαδικασία διεθνής. Και από αυτήν την άποψη υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπό το φως των γεγονότων και η ε, οποία θα ε, πρέπει να ε, συντονίζεται στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ. Ο ΙΚΑΟ αντέδρασε στο δυστύχημα αυτό Μπορούμε να συζητήσουμε γιατί έγινε μετά το δυστύχημα, αλλά είναι σημαντικό για μένα ότι κάθε πρωτοβουλία που θα αναλυφθεί μετά από αυτό το δυστύχημα δεν θα πρέπει να έχει περιφερειακό χαρακτήρα, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την υποστήριξη να το πω έτσι, των ευρωπαϊκών μεταφορών. Αυτό που έκανε η ΙΚΑΟ είναι να δημιουργήσει αυτή την task force προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του συστήματος, η κοινοποίηση των πληροφοριών δηλαδή. Στην παρουσίασή μου είπα ποιες είναι οι ευθύνες ε, των κρατών μελών, αλλά όπως είπε και ο κύριος Μάτιν είναι φανερό ότι κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους για διάφορους λόγους. Ίσως ενδεχομένως ε, να μην έχουν και εκείνα ε, συγκεκριμένες πληροφορίες στη διάθεσή τους ή μπορεί να κρίνουν με σφαλμένο τρόπο κάποιες πληροφορίες που λαμβάνουν. Οπότε, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ΙΚΑΟ είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα. Το να αφήσουμε τις αρμοδιότητες έτσι έχουν σήμερα, το να μην αλλάξουμε τίποτα, να τονίσω ε, ότι ορισμένα μέλη του Συμβουλίου του ΙΚΑΟ ε, πρότειναν και κάποιες τροποποιήσεις της διάσκεψης του Σικάγο, της σύμβασης του Σικάγο. Είναι και πολύ χρονοβόρα αυτή η διαδικασία βέβαια. Γεγονός πάντως είναι ότι ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις ευθύνες όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες, αλλά αν υπάρχουν πληροφορίες βάσει των οποίων θα λάβει κάποιο κράτος μέλος μια απόφαση ή θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν σε άλλο κράτος μέλος, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να εισάγονται σε μια παγκόσμια πλατφόρμα. Αυτός είναι ο στόχος της Task Force που δημιούργησε η ΚΑΟ με στόχο να υποβάλει τις προτάσεις της έως το τέλος ε, του Οκτωβρίου όσον αφορά τη δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας για την ενιαία ανταλλαγή τέτοιου είδους πληροφοριών. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η ενημέρωση των επιβατών. Νομίζω ότι οι σημαντικότερες πληροφορίες που το σύστημα θα πρέπει να δίνει είναι ότι το σύστημα είναι ασφαλές. Και αυτό θα πρέπει να ε, τονιστεί όπως γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής, το 2013 3 δισεκατομμύρια ε, επιβάτες ε, διακινήθηκαν το 2013 με καθόλου ε, θανάτους, με πάρα πολύ λίγους θανάτους, καθόλου θανάτους στην ε, Ευρώπη. Άρα οι δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν θα πρέπει να αναλυφθούν σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορούμε να, ε, κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που θα λέει ότι οι, ε, επιβάτες θα πρέπει να επιλέγουν ε, την, τη διαδρομή. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να, να διασφαλίσει την, τη συνέπεια και την συνοχή του συστήματος. Οι πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται στους επιβάτες είναι ε, ότι το συνολικό σύστημα είναι ασφαλές και αντιμετωπίζει και τα αδύναμα σημεία του. Για το σχόλιο που ακούστηκε και που σχετίζεται με τον συντονισμό στην Ευρώπη και το αν και κατά πόσο υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς στην Ευρώπη, ε, αυτό αποκλείεται. Αυτό δεν ισχύει. Πρώτον, το, σύστημα, το ευρωπαϊκό σύστημα είναι πράγματι περίπλοκο ε, αλλά οι πληροφορίες που εισάγουν οι ευρωπαϊκοί φορείς είναι σαφείς και δεν υπάρχει καμία, κανένας, καμία συσχέτιση του, του δυστυχήματος με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί φορείς. Σταματώ εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο Ζαν Καλό Μπον έχει το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν τέθηκαν συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις προς την ΙΑΤΑ, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές. Η πρώτη αφορά την πολυδιάσπαση και την επικάλυψη, που δεν είναι φίλες αυτές οι δύο έννοιες της ασφάλειας. Το πρόγραμμα Single European Sky είναι ένα από τα προγράμματα τα οποία θα βελτιώσουν το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο βέβαια όπως είπα είναι αρκετά ασφαλές να γίνει ασφαλέστερο γιατί έτσι θα αποφύγουμε τις ε, μη απαραίτητες επικαλύψεις και θα επιτρέψουμε την σωστότερη ανταλλαγή πληροφοριών και διαδικασιών. Υποστηρίζουμε το πρόγραμμα αυτό λοιπόν και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο αυτό σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους νομοθέτες θα μπορέσουν να προχωρήσουν με αρκετή ταχύτητα για να το βελτιώσουμε και να ωφεληθούμε από αυτό. Τώρα για τις αιτίες του ατυχήματος. Για μια ακόμη φορά να πω ότι έχει ξεκινήσει μια επίσημη έρευνα. Η επίσημη αυτή έρευνα της έρευνας ηγείται ε, το Συμβούλιο Αεροπορικής Ασφαλείας των Κάτω Χωρών. Υπάρχει εκπρόσωπος της ΙΚΑΟ. Στόχος της έρευνας αυτής δεν είναι το να κατανείμει ευθύνε, αλλά να κατανοήσει τις αιτίες του ατυχήματος και να αποτρέψει την επανάληψή του. Γι' αυτό λοιπόν στην παρούσα φάση γνωρίζουμε ότι οι έρευνες παρεμποδίζονται λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στο σημείο της πτώσης του αεροσκάφους. Πάντως οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν τις αιτίες του αεροσκάφους και να αποτρέψουν την επανάληψή του. Πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την πλήρη εικόνα του τι έχει συμβεί και να μας δώσουν ε, τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα. Ευχαριστώ. Ο Πατρική έχει το λόγο. Thank you, Mr. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο θέμα και κάτι που είπε ε, ο προλαλής και στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε είναι ότι όντως ένα κράτος είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της ασφάλειας στον αέριο χώρο του και άρα και για την ενημέρωση των αερομεταφορέων και την κοινότητα γενικά σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν στον αέριο χώρο του και για την έκδοση πιθανώς και νόταμ είναι υπεύθυνο το κράτος μέλος. Το κράτος. Αλλά μερικέ φορές τα κράτη μπορεί να μην, να μην κάνουν την ίδια αξιολόγηση του κινδύνου όπως κάποιο άλλος. Για να σα δώσω μόνο ένα παράδειγμα, και αυτό υπάρχει στην ενημέρωση που σα κάναμε, στην περίπτωση της Ουκρανίας. Τον Απρίλιο, όπως ξέρετε, Λόγω της προσάρτησης της Κρυμαίας από τους Ρώσους, η Ρωσία εξέδωσε μία νότα που έλεγε ότι από εδώ και πέρα ο εναέριος χώρος της Κρυμαίας είναι ρωσικός εναέριος χώρος. Και παράλληλα με αυτό, η Ουκρανία είπε «Όχι, είναι ακόμα δικός μας εναέριος χώρος». Και άρα ο κίνδυνος ήταν ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος έμπαινε σε αυτή τη ζώνη δεν θα ήξερε ποιον πύργο κινδύνου, ε, ε, πύργο ε, ενέργεια κυκλοφορία να ρωτήσει. Αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είπαμε στα κράτη-μέλη και στις αεροπορικές εταιρείε, ε, συστήσαμε μάλλον, να μην ε, περνάνε από αυτή την περιοχή. Ε, το, ο διαχειριστής του δικτύου της Eurocontrol εφάρμοσε μέτρα για το κλείσιμο αυτής της περιοχής και η ΆΣΑ δημοσίευσε ένα bulletin που αναφερόταν στις συστάσεις του ΙΚΑΟ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η ΕΑΣΑ ε, ένα μήνα ή δύο μήνες αργότερα έλαβε μία επιστολή από την Ουκρανική Αρχή ε, Πολιτικής Αεροπορίας που έλεγε ότι τώρα μπορούμε να ανοίξουμε κάποιους διαδρόμους μέσα σε αυτόν τον εναέριο χώρο. Η δική μας αξιολόγηση και εκτίμηση ήταν ότι δεν ήταν ακόμα ασφαλής αυτός ο χώρος και γι' αυτό διατηρήσαμε τη σύσταση αυτή ασφαλείας να μην περνάει κανείς από αυτόν τον αέριο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τελικά ο παράγοντας κλειδί είναι οι πληροφορίες, η κοινοποίηση των πληροφοριών και ε, ο χαρακτηρισμός αυτών των πληροφοριών. Εμείς, γιατί ξέρουμε ε, τον τομέα, καταλαβαίνουμε τον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας, καταλαβαίναμε ότι η εκτίμηση που έκανε η Ουκρανία δεν ήταν αναγκαστικά η πιο ασφαλής εκτίμηση υπό τις συνθήκες αυτές. Τις τελευταίες εβδομάδες ακούσαμε πολλές φορές για τη Συρία, τη Λιβύα, το Αφγανιστάν, το Ιράκ αυτές οι χώρες δεν εξέδωσαν καμία νότα που να λέει κλείνουμε τον αέριο χώρο μας γιατί είναι επικίνδυνος. Οι Αμερικάνοι εξέδωσαν νότα προς τις δικές τους αεροπορικές εταιρείες που απαγόρευαν ε, την πτήση ε, πάνω από αυτές τις αυτές για τις Αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες. Ε, καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο λοιπόν και σύνθετο είναι το θέμα. Τελικά πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να γίνεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών στο ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο παγκόσμιο επίπεδο γνωρίζοντας ότι στον ΙΚΑΟ ως μέλη υπάρχουν η Ρωσία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, όλοι τους. Πρόκειται για μια διακυβερνητική οργάνωση όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα ουσιαστικά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι περιορισμοί που υπάρχουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά στην Ευρώπη πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ε, ανταλλαγή πληροφοριών και να ε, καταλαβαίνουμε και το είδος των πληροφοριών, ε, ε, τη φύση των πληροφοριών. Γιατί η ανταλλαγή των πληροφοριών, όπως σας απέδειξα, δεν είναι αρκετή. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι η φύση αυτών των πληροφοριών. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Για την ερώτηση αν υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες, πάρα πολλοί ρόλοι. Όντως υπάρχουν κάποιοι παίκτες. Στα, στην Ευρώπη υπάρχουν 28 κράτη-μέλη, 28 ε, πάροχοι. Ε, αυτό ήδη δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι οι κανόνες, όπως είπε ο Σαλβατόρε, είναι αρκετά σαφείς. Αυτό που μπορεί να ενισχυθεί, πιστεύω, είναι η ροή πληροφοριών μεταξύ όλων αυτών των παικτών στην ε, νομοθετική πρόταση ε, ΣΕΣ 2 ε, ΣΥΝ υπήρχε μία πρόταση για την ευθυγράμμιση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΑΣΑ ούτως ώστε να γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με καλύτερο τρόπο από ό,τι γίνεται σήμερα. Έγινε μία ερώτηση για τα παράσιτα των ραντάρ, τις παρεμβολές. Ε, ε, υπήρξαν κάποια τέτοια φαινόμενα, τα οποία όμως δεν σχετίζονται καθόλου με την περιοχή της Ουκρανίας και αυτό συνέβη ούτως ή άλλως στις αρχές Ιουνίου. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν καθόλου να συσχετιστούν τα δύο γεγονότα. Όσον αφορά το ρόλο μας για την ε, διερεύνηση των ατυχημάτων, αυτό ορίζεται σαφώς στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε παρατηρητές, υποστηρικτές. Εμείς δίνουμε στους ερευνητές της ε, γνώσης και ε, τον σύνδεσμο με την αερονοφυγική βιομηχανία και ε, τη συνεργασία με τα κράτη, ε, μέλη ε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Ολλανδική Ομάδα Έρευνας. Δεν έχουμε δικαίωμα βεβαίως να μοιραστούμε πληροφορίες με κανέναν, εκτός αν αυτή η ομάδα διερεύνηση της Ολλανδίας αποφασίσει η ίδια να κοινοποιήσει τι σχετικέ πληροφορίε. Εμεί δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Τώρα, όσον αφορά τις πιθανές λύσεις, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν χρειάζεται να οικοδομήσουμε συστήματα ε, ευρωπαϊκά πολλών εκατομμυρίων για να έχουμε τουλάχιστον αυτή την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ε, θα πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι διαδικασίες και ποιοι είναι οι οργανισμοί που μπορούν να ε, ανταλλάξουν πληροφορίες εμπιστευτικές ή μη, να χαρακτηριστούν οι πληροφορίες εμπιστευτικές και μη, σε ποιο βαθμό μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τι ε, εμπλοκή θέλουμε εκ μέρους των στρατιωτικών αρχών και αν είναι εφικτό να γίνει αυτό είναι δυνατόν να αρχίσουν οι συζητήσεις με κάποιους ε, στρατιωτικούς φορείς για τα θέματα αυτά. Ε, νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους θεσμούς αυτούς για να υπάρξει αυτός ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος με τα κράτη-μέλη, την Eurocontrol και την EASA. Ε, ε, μεταξύ όλων αυτών θα πρέπει, είμαι σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος να υπάρχει καλύτερη ροή πληροφοριών από ό,τι υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ σύντομα κύριος Μπάλτουιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συζήτηση και ευχαριστώ όλους όσους έθεσαν ερωτήματα. Ε, άκουσα πολλές φορές ε, να ορίσουμε ποιοι είναι υπεύθυνοι. Να το πω σαφώς. Η πρώτη και κύρια ευθύνη για αυτό το τρομερό ε, δυστύχημα βαρύνει εκείνους που εκτόξευσαν πύραυλο σε αεροσκεύος. Αμέσως μετά την ε, ε, κατάρριψη, αυτοί που εκτόξευσαν τον πύραυλο θα πρέπει να ε, περάσουν από δίκη. Είναι, ένα, είναι μια βασική αρχή την οποία δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε έτσι απλά. Όπως είπε και ο, Πάτρικ, είναι πολύ περίπλοκη η περιοχή αυτή, ο, το, ο τομέας αυτός όσον αφορά το πώς τον ρυθμίζουμε και ποιες διατάξεις ισχύουν. Με την ευρύτερη έννοια εμείς οι αρχές και νομίζω ότι ε, εκπροσωπούμαστε πολύ καλά εδώ σε αυτό το πάνελ θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε, πότε το κάνουμε, πώς το κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι είναι σαφές το ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι οι πληροφορίες διανέμονται και κοινοποιούνται σωστό, σωστά, με το σωστό τρόπο και ότι είμαστε αποτελεσματικοί όσο μπορούμε. Όπως είπε και ο Σαλβατόρο και ο Πάτρικ, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες είναι σαφείς, όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να βελτιώσουμε τις ροές πληροφοριών και υπό το φως των συζητήσεων που έχουμε αυτές θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε τις συγκεκριμένε ε, αρμοδιότητες και να προσθέσουμε ή να τροποποιήσουμε τους ρόλους που υπάρχουν προκειμένου να μειώσουμε ή και να εξαφανίσουμε, αν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, τον κίνδυνο να ξανασυμβεί ένα τέτοιο δυστύχημα. Όσον αφορά τη συμμετοχή της Κομισιόν, της ΙΑΣΑ, της, ε, της Eurocontrol στην ε, Task Force του ΙΚΑΟ, αυτό που εξετάζουμε είναι ποιου τομεί, ποια θέματα μπορούμε να βελτιώσουμε. Και ένα τελευταίο πράγμα. Καλό τους πάντες να συνεχίσετε να μας πιέζετε για ε, απαντήσεις. Αλλά σας παρακαλώ μην προτρέχετε να εξάγετε, ε, ε, μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα και μην ακούτε τις θεωρίες συνωμοσία που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Τελευταία πληροφορία που σχετίζεται με τις ε, έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Ολλανδική Αρχή. Ε, βεβαίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο σημείο του δυστυχήματος εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Προτάθηκε ότι η Βρετανική ε, Αρχή Ασφάλειας θα πρέπει να εξετάσει τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και να εκδώσει ένα προκαταρκτικό, ε, μια προκαταρκτική έκθεση. Αλλά όσον αφορά την ευθύνη και τη λογοδοσία, να ε, πω ότι η Ολλανδική Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ποινική δίωξη στη βάση της εθνικής νομοθεσίας, ώστε να ε, προσδιοριστούν οι ευθύνες που ενδεχομένως να βαρύνουν και άτομα και άλλα κράτη. Και ε, η πρώτη ακρόαση έγινε στην Χάγη στις 28 Ιουλίου. Τελευταίο ζήτημα που αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Φυσικά είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που έχει παράσχει το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό το πρόγραμμα και να πω ότι αν είχαμε ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό ε, δεν θα μπορούσαμε πάλι να είχαμε συνολικά εξαφανίσει τον κίνδυνο να συμβαίνουν τέτοια ε, ατυχήματα. Το το δυστύχημα αυτό δεν θα μπορούσε να είχε ε, αποφευχθεί ε, πλήρως στη βάση μόνο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός βεβαίως θα συμβάλλει στην ασφάλεια και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να συσχετίσουμε ε, άμεσα το δυστύχημα με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Προτού δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές, υπάρχει κάποια ερώτηση η οποία δεν απαντήθηκε Παντήθηκε. πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή, γιατί θέλω να, κάνω, να θέσω ένα ζήτημα διαδικαστικό. Ε, έθεσα ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Είπα πώς γίνεται κάποιες αερογραμμές, μεταξύ αυτών και οι British Airways, από τις 14 Ιουλίου δεν πραγματοποιήσουν πτήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Ισχύει καταρχάς αυτή η πληροφορία. Μπορεί κανείς να μην θέλει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, διότι οι έρευνες βρίσκονται σε, ακόμη, σε εξέλιξη. Αλλά το ερώτημά μου είναι αυτό. Υπάρχουν αερογραμμές που είχαν καλύτερες πληροφορίες σε σύγκριση με άλλες και γι' αυτόν τον λόγο δεν πραγματοποιούσαν πτήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν έλαβα απάντηση. Ευχαριστώ ο Ισμαός Χέρτουγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Αλλά για τα ερωτήματα που τέθηκαν, εγώ έθεσα πέντε. Δεν, δεν θα τα επαναλάβω όλα. Ένα όμως που ήταν σημαντικό και δεν απαντήθηκε είναι το εξής. Ρώτησα αν είναι σωστό ότι στις αρχές Ιουλίου υπήρξε μια διαταραχή της ασφάλειας των πτήσεων στις Ανατολικές Άλπεις και μήπως αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο κατέστη αόρατο το αεροσκάφος της πτήσης MH17 ε και ίσως δεν ενημερώθηκαν οι αυστριακές ε, αρχές. Το ξαναλέω διότι αυτή η εξωτερική πηγή διαταραχής ήταν αποτέλεσμα άσκησης του ΝΑΤΟ στην Ουγγαρία. Διότι απενεργοποιήθηκε ένα σημαντικό τμήμα του εξοπλισμού λόγω αυτής της άσκησης. Αυτό είναι σημαντικό ώστε να το γνωρίζουμε στο μέλλον και να μπορούμε να προετοιμαζόμαστε. Ευχαριστώ, κύριε Χαρονίσκο. Uh, uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας θα μου επιτρέψετε όμως να επαναλάβω την ερώτησή μου. Άκουσα κάτι για μια ομάδα, την Task Force, η οποία θα είναι σε θέση να αξιολογεί τις πληροφορίες που συλλέγονται. Και ο κύριος Κι αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών. Και γι' αυτό θέτω το ερώτημά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπεύετε να, κάτι, να κάνετε κάτι άμεσα αξιολογώντας πρώτα βέβαια αυτό το οποίο συμβαίνει, συνέβη. Αυτό σημαίνει ότι θα προτείνεται αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Νομοτεχία. Κύριε Μάιστερ, τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μάθω κύριε Μπρένερ αν έρχεται επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες παίρνετε πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες. Θα έχετε ανάγκη από τέτοιου είδους ε, πληροφορίες. Καλώς ε, σας δίνω το λόγο, ε, ίσως όχι σε όλους, αλλά για να απαντήσετε για τον κύριο Βαντάλ και για την British Airways. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Πατσουκή Πράγματι ε, ήδη υπήρχαν διακοπές στη χρήση των ραντάρ σε μια περιοχή όχι μόνο που καλύπτει την Αυστρία αλλά και οι γειτονικέ χώρες ανάμεσα στις 5 και 10 Ιουνίου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πτήση της ε, Μαλέζιαν ε, που ήταν σε άλλη ημερομηνία και σε διαφορετική κάλυψη ραντάρ. Εμείς τεχνικά ελέγχουμε το τι συνέβη στην περίπτωση αυτή και γιατί διεκόπη η κάλυψη των ραντάρ. Εμείς ε, μιλάμε με τις ε, οργανώσεις οι οποίες είδαν το πώς συνέβησαν οι διακοπές αυτές στην κάλυψη, δηλαδή στην Αυστρία και στις γειτονικές χώρες. Είναι μια τεχνική έρευνα η οποία συνεχίζεται Εξ αρχής είχαμε εμεί κάποιες υποψίες ότι αυτό θα μπορούσε να έχει σχέση με στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά μέχρι τώρα δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό και συνεχίζουμε να αξιολογούμε την κατάσταση σε συνεργασία με την ΆΕΣΑ. Καμία σχέση λοιπόν με την πτήση της Μαλέζια. Διαφορετικές ημερομηνίε, διαφορετική περιφέρεια. Τώρα, για την περίπτωση του θέματος της British Airways, όπως σας είπα, υπάρχουν πολλές επιλογές για να πάει κανείς από το Α στο Β. Η British Airways επέλεξε μια διαφορετική οδό από τη Malaysian, η οποία όμως Malaysian ακολούθησε ένα ανοιχτό δρόμο, όπως το επιβεβαίωσαν και οι Ουκρανικές αρχές. Ε, στην Ευρώπη γίνονται 30.000 πτήσεις την ημέρα και γι' αυτό ακριβώς σας είπα και εγώ και οι συνάδελφοι εδώ ότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής ε, ε, διαδρόμων. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγει κανείς τον ένα ή τον άλλο διάδρομο δεν είναι πάντα γνωστός. Μπορεί να απλά να είναι κάποιες καθυστερήσεις, μπορεί να είναι κάποια άλλα τεχνικά θέματα. Το θέμα τώρα των ε, μυστικών υπηρεσιών είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα όπως ξέρετε. Όπως σας είπα, εν μέρη οι πληροφορίες αυτές μας δίδονται και χρησιμοποιείται. Εν μέρη όμως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί θέμα. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση συνολικά. Και αν εμείς στην Ευρώπη θέλουμε να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα, θα πρέπει να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Με αυτό θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοί μου. Καλώς, σας ευχαριστώ λοιπόν. Ε, οι υπόλοιπες ερωτήσεις. Ποιος θέλει να ξεκινήσει με τις ερωτήσεις. Τρία λεπτά ο καθένας από αυτούς που θα θέσουν τις ερωτήσεις. Μπαρ. Sorry. Ε, ε, ναι. Mr. Bach says ladies first. Ms. Foster, then we can discuss now half an hour or one hour about who is uh, talking. Come on, yeah. Sorry, I missed. Εσείς λοιπόν. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων και της Κομισιόν που ήρθαν εδώ σήμερα. δεν θα μπορούσα να τα πω πιο εύγλωτα από ό,τι τα είπε ο συνάδελφος Βαντάλεν, τις τραγικές συνέπειες δηλαδή ε, μιας τέτοιας ε, τρομοκρατικής ενέργειας. Και ε, για να πάω λίγο πιο πίσω, ε, οι αρωματαφορές ήταν ο κλάδος μου, ίσως ε, ε ξέρετε κάποιοι από εσά. Πέρασα τη μισή ζωή μου σε ύψος 35.000 ποδιών και κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο έχεις ε, απολύτη εμπιστοσύνη ε, στις ε, ε, κρατικές υπηρεσίες, ε, ε, σε όλο το σύστημα που υπάρχει. Είναι ένα από τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς. Αλλά θυμάμαστε στο Λόκερμπι το πλάνο το 474 γιατί κάποιος έβαλε εκρηκτικά μέσα στην πτήση και τώρα μιλάμε για το ατύχημα αυτό των μαλισσινών αερογραμμών. Προσπαθούμε να βρούμε μέσω της νομοθεσίας ε, ε, τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας των μεταφορών. Αλλά πριν από μερικά χρόνια είχαμε την, ε, την 11η Σεπτεμβρίου. υπάρχουν καμικάζι που ε, ε, σκοτώνονται στην προσπάθεια της τρομοκρατικής ε, επίθεσης. Και όλο αυτό μας οδήγησε στο να ξαναδούμε τα μέτρα ασφάλειας στα αεροδρόμια και να αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνδυνο. Ήταν μεγάλο το τίμημα. Και τώρα προχωρούμε στο τελευταίο αυτό επεισόδιο. Γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να το προβλέψει εκ των υστέρων. Είναι εύκολο να πει κανείς ε, και να ρίξει τις ευθύνες. Αλλά δεν μπορεί να το προβλέψει. Νομίζω ότι την ευθύνη την έχουν αποκλειστικά οι Ρώσοι, η ρωσική κυβέρνηση. Ε, μπορούμε βέβαια να απευθύνουμε κατηγορίες δεξιά και αριστερά, αλλά αυτό ε, δεν μας οδηγεί πουθενά. Αυτοί και μόνο έχουν την ευθύνη. πιστεύω ότι έγιναν λάθη όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους και τα σχέδια πτήσης κατά τη γνώμη μου. γιατί ε, δεν ήταν ε, μόνο οι Μαλισσιανές αερογραμμές, οι Virgin, οι KLM ακολουθούσαν ε, τον ίδιο αεροδιάδρομο. Αν έρθουμε λοιπόν στη σημερινή στιγμή, το ερώτημα είναι τι θέλουμε να βγάλουμε από αυτή την ακρόαση. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και νομίζω ότι υπάρχουν δύο ερωτήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και πιστεύω ότι θα έχουν την υποστήριξη της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου. Το ένα αφορά την επικοινωνία, όπως είπατε, βασιζόμαστε πάρα πολύ σε πληροφορίες στρατιωτικές και πολιτικές ε, και είπατε ότι ε, θα μπορούσε να βελτιωθεί ε, το θέμα αυτό και έχει την υποστήριξή μας και σε, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Και τέλος, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και το ΣΕΖΑΡ, για να γίνουν αυτά χρειάζεται περισσότερη πολιτική βούληση. Ε, να είμαστε όλοι μαζί για τα θέματα αυτά και όχι ο καθένας χωριστά. Και το ίδιο ισχύει και με το ΣΕΖΑΡ ε, που θα βελτιώσει συστήματα ε, επίγεια και αέρια... Αυτά ήταν κάποια σχόλια που ήθελα να κάνω και πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά όλους αυτούς τους κυρίους που ήρθαν σήμερα να μας εξηγήσουν ποιος είναι ο ρόλος τους και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα συμπεράσματα της κυρίας Φώστερ. Ήταν ιδιαίτερως διαφωτιστική η συγκεκριμένη ακρόαση. Πολύτιμη θα έλεγα. Τώρα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις ζώνες κρίση στο μέλλον. Είπαμε ότι οι πληροφορίες συλλέγονται και προέρχονται από τα κράτη-μέλη συνήθως. Τι μπορούμε λοιπόν εμείς, ε, με ποιο τρόπο μπορούμε ε, σοβαρά να σκεφτούμε ότι τα κράτη-μέλη συλλέγουν αποκλειστικά αξιόπιστες πληροφορίες. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές είναι χαοτική. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το να γνωρίζει κανείς ε, το ποιος αξιολογεί την ποιότητα της πληροφορίας. Τώρα η αξιολόγηση του κινδύνου, το επίπεδο, του επίπεδου του κινδύνου. Εάν κριθεί ότι είναι αποδεκτή ή αποδεκτό το επίπεδο τότε δίδεται η άδεια για την ε, τέλεση της πτήσης. Αλλά ε, για κάποιον το αποδεκτό μπορεί να είναι για άλλον το απαράδεκτο. Συνεπώς υπάρχουν και τα οικονομικά τα οποία ε, παίζουν κάποιο ρόλο. Θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη πλέον ερώτηση. Μας είπατε ότι δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε παρά μόνο συστάσεις. Πρόκειται για δεσμευτικές συστάσεις. Ε, δεν πρόκειται για απαγορεύσεις, δεν έχουν άμεση εκτελές, δεν εκτελούνται άμεσα. Σε ποιο βαθμό γίνονται σεβαστές αυτές οι ανακοινώσεις. Ευχαριστώ κύριε Σπρινσκή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα σημείο, σε ένα ζήτημα γενικής φύσεως. Ακούστηκε ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των πτήσεων βαρύνει τα επιμέρους κράτη. Ταυτόχρονα όμως ακούμε εκκλήσεις να προχωρήσουμε στη δημιουργία των ε, στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανή που ε, σηματοδοτεί μια μεγαλύτερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και μια προσδοκία ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού μπορούμε να διασφαλίσουμε με καλύτερο τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπόλβιν και τους άλλους να εξετάσουν αν υπάρχει ανάγκη να επανεξεταστεί προσεκτικά η πρόταση, οι προτάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο της ε, πρωτοβουλίας του ΠΛΑΣ που αφορούν και την εναρμόνιση των, ε, ε, του κανονιστικού πλαισίου και τον, ε, το καθεστώς που διέπει την EASA. Καταλαώ ότι η επιχειρηματολογία που έχει προέλθει από την Κομισιόν είναι ότι ε, όλα αυτά γίνονται για τον εξορθολογισμό του συστήματος κτλ. Στην ε, πρωτοβουλία, δεύτερο ερώτημα, στην πρωτοβουλία που αφορά αυτή την, την ασφάλεια των πτήσεων, ίσως θα πρέπει να ε, ε υιοθετηθεί και μια άλλη ε, προσέγγιση. Η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας θα πρέπει να διαχωριστεί σε επιχειρησιακό κομμάτι και σε υποστηρικτικό κομμάτι, με πιθανότητα να υπάρξει και ε, ιδιωτικοποίηση των δραστηριοτήτων υποστήριξης υπάρχει και μια ε, προσέγγιση που κατατείνει στην συγκεντροποίηση του δικτύου του συστήματος ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Αυτό που θέλω να θέσω είναι η ανάγκη να ε, υπερισχύσει η ανάγκη διασφάλισης ασφάλειας των πτήσεων έναντι άλλων κριτηρίων. Για παράδειγμα, οικονομική βιωσιμότητα, αποδοτικότητα, ο εξορθολογισμός του συστήματος που έχουν όντως και εκείνα μία χρησιμότητα, αναμφισβήτητα, αλλά όπως είπε και ο κύριος Σακητάνου, το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο σε τελική ανάλυση Οπότε, αυτό που θα πρέπει να κυριαρχεί στη σκέψη μας είναι να υπάρχει καλύτερο σύστημα κοινοποίησης πληροφοριών, να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες που ενδεχομένως υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά χωρίς να θυσιάσουμε για το σκοπό αυτό την ασφάλεια. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Άντερσον. Κύριε Άντερσον. Πρώτα απ' όλα να υποστηρίξω τα ερωτήματα και τα σχόλια που ε, ακούστηκαν από τους συντονιστές και τους συναδέλφους. Εγώ πρέπει να σας πω ότι νιώθω ότι δεν λάβαμε απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που θέσαμε. Οπότε θα ήθελα να συνοψίσω και να ξανατονίσω ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα. Σε τελική ανάλυση δεν μας βοηθά το γεγονός ότι ε, να, λέμε ότι η ευθύνη βαρύνει τους ε, ε, αυτονομιστές. Διότι αν ε, υπήρξε παραβίαση της Σύμβασης του Σικάγο λόγω συγκεκριμένων ατόμων και συγκεκριμένων κρατών μελών ή άλλων κρατών που γνώριζαν πληροφορίες αλλά δεν τις κοινοποίησαν, τότε αυτό χρειάζεται ε, διερεύνηση. Αλλά δεν χρειάζεται να μας πείτε ότι είναι οι αυτονομιστές εκείνοι που ευθύνονται. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, ήταν γνωστό ότι οι αυτονομιστές είχαν στη διάθεση του τέτοιον στρατιωτικό εξοπλισμό και γι' αυτό το λόγο όσον αφορά το ερώτημα που σχετίζεται με την British Airways έχω ένα ερώτημα προς την Eurocontrol και, και άλλους. Μιλήσατε με την British Airways για, το, για ποιον λόγο λάβαν την απόφαση που έλαβαν διότι υπάρχουν νομικά ζητήματα, ζητήματα που σχετίζονται με τη λογοδοσία και είναι πολύ καλό το ότι ήρθατε εδώ και μας μιλάτε, αλλά νιώθω ότι δεν λαμβάνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Και δεύτερο συγκεκριμένο ερώτημα για την τεχνολογία. Θέλω να μας πείτε ποιες ξεχωριστές ανεξάρτητες τεχνολογίες ε, ε, και για τη δημιουργία ποιων τεχνολογιών ε, χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Πρόγραμμα ώστε να μην βασιζόμαστε σε ε, στρατιωτικές ε, πληροφορίες. Και τρίτον, δεν με ικανοποιεί η απάντηση για την ενημέρωση των επιβατών. Φυσικά κατανοώ ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τους επιβάτες, αλλά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε δίκιο όταν είπε ότι υπάρχει και μια ε, πιθανότητα να αλλάξει το πρόγραμμα πτήση, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην ενημερώνουμε τους επιβάτες για το ποια θα είναι η πτήση που θα ακολουθηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω για άλλη μια φορά τα συλληπιτήριά μου σε όλους όσοι με τον ένα τον άλλο τρόπο ενεπλάξαν σε αυτό το δυστύχημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέλη. Ε, Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε λεπτομερείς παρουσιάσεις των διαδικασιών που ακολουθούνται στον τομέα της ασφάλειας των πτήσεων, της ανταλλαγής πληροφοριών, στο πρώτο τμήμα της ακρόασης. Είναι προφανές ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή αυτών των μηχανισμών. Ειδικά στην τραγική αυτή περίπτωση του Μαλαισιανού αεροσκάφους. Φυσικά και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών είναι κομβική. Φυσικά και αυτοί οι οποίοι κατέριψαν το αεροσκάφος θα πρέπει να δικαστούν και το είπατε αυτό, αλλά τίθεται σαφώς και το θέμα των κρατών μελών που συμμετέχουν στις διεθνείς οργανώσεις που δίδουν τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται. Οι διεθνείς οργανώσεις έχουν συνήθως τους δικούς τους κανόνες και τις δικές τους διαδικασίες σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Αν δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους, που προέρχονται από τα κράτη-μέλη και όπως υπόθηκε ήδη υπάρχει και θέμα σχετικό με την αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών που προέρχονται από τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ε, και αυτοί τα δικά τους προβλήματα γιατί αντιπροσωπεύουν ε, περιοχές κρίσης στην παρούσα φάση. Θα ήθελα να μάθω και τι γίνεται με τους εσωτερικούς μηχανισμούς τους οποίους ενεργοποιείται όταν κάποιες χώρες πιθανώς δεν εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους όπως θα έπρεπε ή εάν οι πληροφορίες, τους, οι πληροφορίες τις οποίες δίδουν δεν είναι τόσο αξιόπιστες όσο θα έπρεπε. και στο ενημερωτικό υλικό το οποίο μας έστειλε η ΑΣΑ στην τρίτη σελίδα λέγεται ότι την 1η Ιουλίου οι υπηρεσίες ε, ελέγχου εναερίου χώρου της Ουκρανίας δημοσίευσαν μια νότα και η ΆΣΑ δεν είχε πάρει την ενημέρωση αυτή πριν από την, ε, από την πτώση του αεροσκάφους που συνέβη στις 17 Ιουλίου. Το θέμα είναι λοιπόν γιατί συνέβη αυτό. και ποιος είναι υπεύθυνος για τη μη λήψη της νότα αυτής. Ευχαριστώ κύριος Ρόμπερτ Ζήλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν εδώ. Νομίζω ότι ο στόχος της συνάντησής μας σήμερα εδώ ήταν ότι πρέπει να δώσουμε και στους οργανισμούς αυτούς κάποιες πολιτικές ε, ε, θέσεις από τη δική μας πλευρά και κάποιες νέες προτάσεις που θα πρέπει να τεκμηριώνονται και με ε, λόγους επαγγελματισμού. Δεν χρειαζόμαστε δεν χρειάζεται πάντοτε να συζητούμε την ζώνη συγκρούσεων. Νομίζω ότι όμως υπάρχει ένα νέο είδος ε, ζώνης συγκρούσεων εδώ στην ε, Ανατολική Ουκρανία, γιατί όπως είπε η Ρωσία πρόκειται για ένα συνδυασμένο πόλεμο. Αν δείτε τις πτήσεις, μπορείτε να, μπορούν να πραγματοποιούνται και κάποιες ε, πτήσεις πάνω από την Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, οπότε υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνονται πτήσεις εκεί από ε, άποψη ασφάλειας, αλλά εδώ στην Ανατολική Ουκρανία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν νέε προσεγγίσει από την ε, πλευρά της Ρωσίας και μια σειρά από κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα σύμφωνα με τον ΙΚΑΟ. Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν μπορεί κανεί να ελέγξει μια περιοχή που είναι εμπόλεμη και που ε, αυτό ε, αφορά και τη νέα προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Ρωσία Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυμβεί. Γιατί, διότι αποκρύπτονται πληροφορίες, αποκρύπτονται πληροφορίες αφενός και αφετέρου ε, δίνονται ε, πύραυλοι στους αυτονομιστές. Όταν λοιπόν η ε, Ολλανδική Επιτροπή καταλήξει τα πορίσματά της, θα πρόκειται για ένα πολιτικό αποτέλεσμα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβιώσει πολιτικά σε αυτή τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και το ζήτημα δεν είναι απλώς ποιος πάτησε το κουμπί για να εκτοξευθεί ε, ένας πύραυλος. Το ζήτημα είναι ποιος επέτρεψε οι αυτονομιστές να αποκτήσουν τέτοιου είδους πυράβλους. Και με αυτό ερχόμαστε και στο δεύτερο επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ολλανδοί συγκεκριμένα πολίτες μετά από αυτό το δυστύχημα δεν θα έχουν καμία εμπιστοσύνη στα, στο σύστημά μας και στους μηχανισμούς μας. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι και να πω κάποια λόγια ακόμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη στη συγκεκριμένη περιοχή την εμπόλεμη. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε στο εξής, ότι κάθε αρχή που θα ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να ενημερώνει τις ε, αερογραμμές και τις αρχές άμεσα. Προφανώς απεκρίβησαν πληροφορίες στη συγκεκριμένη περίπτωση και ε, η προσέγγιση που υιοθετήθηκε ήταν ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τη συγκεκριμένη περιοχή και αυτό ήταν τραγικό. Ε, ειδικά για τους ανθρώπους που είχαν συγγενείς και φίλους στη συγκεκριμένη πτήση. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε και να υιοθετήσουμε μια ε, νέα προσέγγιση. Για, την, για τις διασυμβηρικές πτήσεις που ε, παραβιάζουν την ε, διάσκεψη του Σικάγου. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί αυτοί οι νέοι κανόνες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν απαγορεύονται οι υπερπτήσεις. Υπάρχει όμως κάποια αντίδραση στην εξέλιξη αυτή από τους εμπειρογνώμονες μας. Ευχαριστώ, ο κ. Ντεγκράντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν πάρα πολλές πληροφορίες. Δεν ήταν και εύκολο πράγμα. Όλοι εδώ σκεφτόμαστε με βάση δύο κεντρικές ιδέες. Την ασφάλεια και την υπευθυνότητα. Ε, για την ασφάλεια προχωρούμε όσο το δυνατόν ε, καλύτερα, στο μέτρο του δυνατού. Ε, αλλά στο θέμα της ευθύνης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, ιδίως σε εμπόλεμες συνθήκες. Πάντοτε λέμε ότι το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια. Ε, εξάλλου, ε, πάντοτε ε, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος ωφελείται από το έγκλημα. Ποιον ωφελεί αυτό το ε, συμβάν. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες θυμάτων. Υπάρχουν τα ανθρώπινα θύματα και μετά υπάρχει και μια αεροπορική εταιρεία. Πρέπει να το πούμε και αυτό μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες είναι πιθανό να εξαφανιστεί εντελώς από το χάρτη η αεροπορική αυτή εταιρεία. Ε, ενώ δεν είναι καθόλου υπεύθυνη για ό,τι συνέβη. Πρέπει να πούμε λοιπόν την αλήθεια. Υπάρχουν ε, πολιτικές θέσεις, υπάρχουν πολύ μεγάλες συζητήσεις που γίνονται επ' αυτού δεν πρόκειται για μια σύγκρουση ίσονος σημασίας. Ε, είναι μια πυρήτη αποθήκη αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία που απειλεί το status quo. Λοιπόν, όσον αφορά τις ευθύνε, το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό έχουμε αρκετά στοιχεία. Έχουμε μια αεροπορική εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίε ε, του ατυχήματος. Ε, υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες θυμάτων που δεν μπόρεσαν να βρουν ε, τη σωρό των συγγενών τους. Ήδη ε, σε κανονικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να ε, προσδιοριστούν οι ευθύνε. και υπό τις σημερινές συνθήκες είναι αδύνατο να υπολογίσει κανείς πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να διερευνηθεί η υπόθεση. Και απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να κάνουμε προτάσεις. Θα πρέπει κάθε εταιρεία να αναγνωρίσει τις ευθύνες της. Τα θύματα αυτά θα είναι θύματα, διπλά θύματα κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός που θα έχει βαρύτατες συνέπειες. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν οι άμεσες ευθύνε. Υπάρχουν ε, φυσικά και όλες οι ζημίες που έχουν προκληθεί ε, σε άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πώς τελικά θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη ε, απέναντι σε αυτή την κατάσταση και τον πόλεμο που κινδυνεύει να επεκταθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για, την, για όλες τις εξηγήσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί για τους διάφορους ρόλους. Ε, η ερώτηση όμως είναι τι διατάξεις, τι μέτρα έχετε λάβει για την πρόσφατη ε, ιστορία με το ηφαίστειο της ε, Ισλανδίας. Είστε προετοιμασμένοι για ενδεχομένη έκρηξη του ηφαίστειου αυτού, γιατί σε προηγούμενες περιπτώσεις ανάλογες ε, ε, είχε το Ηνωμένο Βασίλειο μεγάλα προβλήματα. Έχω και εγώ μια ερώτηση που αφορά πάντοτε την εθνική κυριαρχία. Η ΦΑΠΣ αποφάσισε ε, ε, αποφασίστηκε πέρσι ε, διότι όμως κάποια κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν το συγκεκριμένο νόμο διότι είναι δική τους αρμοδιότητα θεωρούν. Όμως θα πρέπει να έχουμε κοινή θέση το καλύτερο θα ήταν ε, παγκόσμια θέση, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Αν το δυστύχημα, το δυστύχημα λοιπόν θα οδηγήσει τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουμε μια κοινή θέση που θα λέει ότι είτε επιτρέπεται είτε απαγορεύονται οι πτήσεις σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή και όχι να, το, να πετούν και οι δε να μην πετούν διότι υπάρχουν και ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος, με την κυροζήνη κτλ. Αν κάποιο κράτος λοιπόν πει ότι απαγορεύονται οι πτήσεις πάνω από τον αέριο χώρο μου, ε, υπάρχουν και κόστη για το κράτος αυτό, διότι δεν καταβάλλονται τέλη. Αν τώρα κάποιοι φορείς λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό, άλλοι λένε ότι μας ενδιαφέρει, υπάρχει και μια στρέβλωση του ανταγωνισμού. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει κοινή θέση, να ενημερωθεί και η κοινή γνώμη και πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, διότι είπατε ότι αυτή είναι η κατάσταση, το κράτος μέλος έχει την ευθύνη του. Για μένα είναι σαφές, πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση η οποία θα υιοθετείται και θα τηρείται από όλα τα κράτη-μέλη ώστε ο ΙΚΑΟ να έχει την, ε, τη δικαιοδοσία να πει ότι εδώ επιτρέπονται οι πτήσεις και εδώ απαγορεύονται οι πτήσεις. Ωραία, και τώρα να κάνουμε έναν τελικό ε, κύκλο απαντήσεων. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, ο κύριος Μπρένερ. Ε, σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση για το Ισλανδικό ηφαίστειο. Η κατάσταση που είχαμε δει όταν είχε εκραγεί το προηγούμενο ηφαίστειο δεν ήταν πολύ ευχάριστη. Ε, πολλά μέτρα έχουν ληφθεί από τότε. Ένα από αυτά είναι η δημιουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων έτσι ώστε ε, να υπάρξει σωστή ανταλλαγή πληροφοριών και των επιλογών που είναι διαθέσιμες. Γιατί κάθε μία από αυτές τις κρίσεις είναι διαφορετική. Η ACCC τις τελευταίες εβδομάδες έχει κινητοποιηθεί δυστυχώς ε, έμπολα, TCM 17 και άλλα θέματα. Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια των δομών που έχουν δημιουργηθεί και των ολοένα πιο εναρμονισμένων διαδικασιών μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε ε, την κατάσταση της ε, μόλυνσης των ουρανών από στάχτη. Δεν θα βιώσουμε αυτό που είχαμε βιώσει στο παρελθόν ε, γιατί τότε είχε δημιουργηθεί αρκετή σύγχυση και πολλά προβλήματα. Οι διαδικασίες λοιπόν στα κράτη-μέλη έχουν όπως είπα ευθυγραμμιστεί και οι συντονισμοί, οι μορφές συντονισμού έχουν ε, πλέον τεθεί σε λειτουργία. Νομίζω ότι είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και θα αποφύγουμε τα επιπτώσεις ε, της προηγούμενης περίπτωσης. Τώρα, για την κατάσταση της υποχρέωσης των κρατών μελών Πράγματι ε, τα κράτη-μέλη κάνουν εκτιμήσεις κινδύνου και αξιολογήσεις κινδύνου για το δικό τους ενέριο χώρο και την ασφάλεια του εθνικού τους κοινού και μέσω του συστήματος NOTAMS να ενημερώνουν. Αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς είναι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη των 28 και το Κοινοβούλιο να σκεφτεί αν πρέπει στο μέλλον να ενθαρρυνθούν όχι μόνο να κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις κινδύνου τις οποίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν, αλλά να μοιράζονται υποχρεωτικά τις πληροφορίες αυτές. Γιατί τότε μόνο, όπως το Eurocontrol, ο manager του δικτύου δηλαδή, θα μπορεί να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες και θα ελέγχει αν οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι συμβατές ή θα πρέπει να υπάρξουν άλλες αποφάσεις ε, που θα ανοίξουν συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Γιατί αν δεν έχουμε τις πληροφορίες δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε στις συζητήσεις λοιπόν. Δεν ξέρω αν η Ευρώπη των 28 μπορεί να, να συμμεριστεί μαζί μας περισσότερες πληροφορίες και στα πλαίσια της συνεργασίας της ΕΑΣΑ και στα πλαίσια της εργασίας με την ΕΚΑΚ γιατί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν υπάρξει κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε μια δεύτερη φάση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρουμε ότι οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, δεν είναι στην Ευρώπη των 28 βέβαια, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Σαλβατόρε Σακιτάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι είστε σε θέση να προφέρετε σωστά το όνομά Να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κύριος Μπριέι. Πρώτον, γιατί η British Airways άλλαξε τις ε, ε, πτήσεις της. Είναι συμβατό με την νομοθεσία κάτι τέτοιο. Η πρώτη και κύρια ευθύνη βαρύνει το κράτος μέλος, αλλά κάθε κράτος μέλος που έχει άλλες πληροφορίες μπορεί να εκδώσει νόταμ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν εκδόθηκε νόταμ, αλλά σύσταση προς την BA να ε, αλλάξει το flight plan. Επρόκειται για μυστική πληροφορία, για στρατητική πληροφορία και αυτό είναι το ζήτημα που συζητούμε στο ΙΚΑΟ. Αυτές, αυτού του είδους θα πρέπει να κοινοποιούνται ώστε όλα τα κράτη-μέλη και οι αερογρομές να μπορούν να λαμβάνουν παρόμοιες αποφάσεις. Φυσικά, το, οι πτήσεις σε εμπόλεμες ζώνες και οι υπερπτήσεις σχετίζονται με τις μυστικές πληροφορίες και τις στρατιωτικές ε, πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην εκάστοτε περιοχή. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα ερώτημα. Ποια είναι η διαχείριση που θα πρέπει να γίνεται όταν ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ε, ε εκτελέσει τις ε, υποχρεώσεις του. Και εδώ πάλι θα πρέπει να κοινοποιούνται οι πληροφορίε ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη. Και αυτό είναι το καθήκον που εξετάζει η Task Force της ΙΚΑΟ. Όσον αφορά μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πτήσεις, ναι, είναι κάτι που χρειάζεται και είναι απαραίτητο. Αλλά και πάλι η πολιτική αεροπορία είναι ένα διεθνές φαινόμενο και οι μαλισσινές αερογραμμές δεν είναι ευρωπαϊκές. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό μηχανισμός ο οποίος ε, ωστόσο θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο ε, μιας παγκόσμιας διεθνούς υποχρέωσης κοινοποίησης πληροφοριών. Όσον αφορά την πρόσβαση στην λήψη απόφασης, είναι σίγουρο ότι όταν υπάρχει διαστήριο, ένα δυστύχημα. Η σύμβαση του Σικάγο ορίζει υποχρέωση να, υπάρχει, να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο σημείο του δυστυχήματος ώστε να διεξαχθούν οι απαραίτητες ε, έρευνες. Δυστυχώς η κατάσταση για την οποία ε, μιλούμε δεν εμπίπτει στον έλεγχο κανενός κράτους μέλους που συμμετέχει στη συγκεκριμένη σύμβαση διότι η περιοχή ελέγχεται από τους αυτονομιστές και αυτό δυσκολεύει βεβαίω την πρόσβαση στη συγκεκριμένη ζώνη. Για τις διασυμβηρικέ πτήσει είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα είναι βεβαίω και πολιτικές, αλλά από άποψη αεροπορίε θα πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση του κανονισμού του Σικάγου. Και υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες δυστυχώς είναι χρονοβόρες σύμφωνα με το άρθρο 84 του, της, διάσκεψης, του, της Σύμβασης του Σικάγου. Η διαδικασία αυτή δεν πρόκειται να μας οδηγήσει σε άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ, ο Ζαν Κάρλο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. Το πρώτο σχετίζεται με την αξιολόγηση του κινδύνου. Και θα ήθελα να τονίσω ακόμη μια φορά, όπως έκανα και στην παρουσίασή μου, ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση κινδύνου, ανεξάρτητα από το πόσο καλά γίνεται, εξαρτάται από την ποιότητα των πληροφοριών στην οποία βασίζεται. Αν έχουμε αξιόπιστες ακριβείς πληροφορίες, τότε μπορούμε να έχουμε μια καλή εκτίμηση του κινδύνου. Διαφορετικά το όλο εγχείρημα δεν είναι, θα έλεγα ότι είναι χάσιμο χρόνο, αλλά η αξία του είναι περιορισμένη πάντως. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ακόμα μια φορά αυτό που είπε ο κύριος Κι. Και ο χαρακτηρισμός των πληροφοριών δεν είναι μόνο το θέμα να έχουμε τις πληροφορίες, αλλά να προσδιορίζουμε ε, τις πληροφορίες αυτές και να καταλαβαίνουμε τι έχει σχέση και τι είναι σημαντικό με την ασφάλεια της πτήσης. Ε, το δεύτερο θέμα αφορά την πληροφόρηση των ε, ε, επιβατών. Όλοι ξέρετε ότι σε τακτικούς ε, επιβάτες δεν κρύβουμε τέτοιες πληροφορίες. Μπορεί κανείς να κοιτάξει τον χάρτη και να δει ε, ποια ακριβώς θα είναι η διαδρομή που θα ακολουθεί δεν κρύβουμε τέτοιες πληροφορίες. Θεωρούμε ότι είναι πληροφορίες που είναι σημαντικό να παρέχονται. Όμως, σε στρατηγικό επίπεδο υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτό. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με την ασφάλεια και πάλι. Σίγουρα δεν θέλουμε άνθρωποι που έχουν άλλα συμφέροντα να ξέρουν ανα πάσα στιγμή που είναι τα αεροσκάφη. Δεν θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των τρομοκρατών πιο πολύ από ό,τι είναι η διεύκολη σήμερα. Και δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα σχέδιο πτήση ε, μπορεί να αλλάξει και να αλλάξει σημαντικά σε τακτικό επίπεδο. Ε, όταν παίρνει το ελεύθερο, μάλλον το, το OK, το τελευταίο, το παίρνει ε, η πτήση μετά το κλείσιμο των θυρών. Ε, ή και τη διάρκεια της πτήσης. Μπορεί ο πιλότος να θέλει να αποφύγει ε, μια θύελα, μια καταιγίδα μέσα στην ε, τροπική ζώνη. Μου συνέβη ε, εμένα όταν ήμουν πιλότος και θα, πρέπει να περάσω από πολλές διαφορετικές χώρες για να το κάνω αυτό. Αυτό είναι τακτική ελιγμή που είναι αδύνατο και συγγνώμη που το λέω να κοινοποιηθούν όλα αυτά εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. και μία ερώτηση για τις συστάσεις στον τομέα της ασφάλειας και σε ποιο βαθμό είναι δεσμευτικές οι συστάσεις της ΑΕΣΑ. Όχι, είναι συστάσεις, συνεπώς όχι δεσμευτικές. Εμείς κάναμε συστάσεις για να σταματήσουν οι πτήσεις στο Τελαβίβ. Ακολουθήθηκε η σύσταση αυτή από όλες τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες εκτός από μία. Οι συστάσεις αυτές δεν είναι μεν υποχρεωτικές, αλλά νομίζω ότι ε, υποχρεώνει αυτούς που δεν εφαρμόζουν τη σύσταση να κάνουν αυστηρότερες αξιολογήσεις κινδύνου και να υποχρεωθούν να τεκμηριώσουν γιατί δεν πρέπει να ακολουθήσουν τη σύσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ενισχύει τις δυνατότητες των συστάσεων της ΕΑΣΑ. Τώρα οι ερωτήσεις για τα νόταμς και γιατί δεν πήραμε νόταμς. Εμείς δεν παίρνουμε τα νόταμς, εμείς δεν είμαστε λειτουργική υπηρεσία. Υπάρχουν χιλιάδες νόταμς οι οποίες ανταλλάσσονται κάθε μέρα στον κόσμο και εμείς δεν είμαστε επιχειρησιακή θα έλεγα υπηρεσία που να τις παίρνει καθημερινά. Αντίθετα όμως ε, κάθε τρεις μήνες ή κάθε έξι μήνες ε, και σε ετήσια βάση όταν υπάρχει μία νότα η οποία κλείνει ένα μεγάλο τμήμα του εναερίου χώρου για λόγους ασφαλείας ε, προφανώς ενημερωνόμεθα και αυτό θα το βελτιώσουμε στο μέλλον. Τώρα για ποιες εταιρείες επιλέγουν να περάσουν πάνω από ποιες περιοχές. Να πάρω ένα άλλο παράδειγμα, το Αφγανιστάν. Για το Αφγανιστάν γνωρίζουμε ότι είναι πόλεμη ζώνη. Γνωρίζουμε ότι γίνονται οι υπερπτήσεις εδώ και χρόνια άνωθεν ε, του Αφγανιστάν. Να σας παραπέμψω όμως αυτό το οποίο είπε ο κυρία Φώστερ και ο κύριο Τσίλε, ότι μιλάμε για νέα είδη απειλών. Υπό το φως δηλαδή αυτών των νέου τύπου απειλών απαιτείται να επανεξετάσουμε το αν η υπέπτυση του Αφγανιστάν είναι ασφαλής. Γιατί γνωρίζουμε τώρα ότι οι τρομοκράτες μετά από αυτό που έγινε στην Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα για να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Πρέπει λοιπόν να το δούμε με διαφορετικό τρόπο και να βρούμε ένα νέο υπόδειγμα αντίδρασης. Τώρα για το Αφγανιστάν, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε απαγόρευσε τι επιχειρήσεις της αεροπορικές της Αμερικανικές να το κάνουν, να πετούν πάνω από τη χώρα. Εμείς ανά εσά στείλαμε την ενημέρωση αυτή σε όλες τις χώρες και σε όλους τους Ευρωπαίους ε, αερομεταφορείς. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να απαγορεύσουμε. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα συλλογής πληροφοριών που θα μας δώσει τη δυνατότητα να πούμε ότι ο κίνδυνος είναι υψηλότατος στο Αφγανιστάν. Οπότε σας συστήνουμε ε, σαφώς να αποφύγετε τον εναέριο χώρο, τον Αφγανικό. Αυτό το οποίο είπαμε όμως είναι ότι οι Αμερικανοί απαγόρευσαν στους αερομεταφορείς τους να πηγαίνουν στη χώρα αυτή ε, εσείς ε, χώρες μέλη, εσείς αερομεταφορείς, εσείς θα αποφασίσετε αν ε, είναι ασφαλές ή όχι να πάτε στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό βέβαια. Θα πρέπει να βρούμε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου εμείς θα μπορέσουμε να εξετάσουμε ποιοτικά τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Δεν θα πρέπει εμείς στην Ευρώπη νομίζω να ακολουθήσουμε τυφλά όλες τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται να προσπαθήσουμε να διαμορφώνουμε και τις δικές μας απόψεις και αντιλήψεις πάνω σε αυτά. Κύριε Βάλβιν, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά να πω ότι είναι πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή και υποψιάζομαι ότι δεν είναι η τελευταία φορά που συζητούμε τα ζητήματα αυτά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και ελπίζω να ξανακαλέσουμε και την Επιτροπή για να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Να δώσω κάποια, ε, ε κάποιες απαντήσεις. Ένα ζήτημα που αφορά ε, την παρεμβολή στα ραντάρ το φαινόμενο, το γεγονός αυτό που έγινε τον Ιούνιο. Συμφωνώ ότι δεν πρόκειται για παράγοντα που συνετέλεσε, αλλά στην Επιτροπή ε, δώσαμε εντολή στην ΕΕΑΣΑ να διερευνήσει το συγκεκριμένο περιστατικό και οι εργασίες αυτές βρίσκονται σε ε, εξέλιξη. Ο κύριος Μαρινέσκου και εσείς κύριε Πρόεδρε, ε, ρωτήσατε αν η Κομισιόν είναι έτοιμη να παρουσιάσει κάποια νέο κανονισμό ε, για τους τομείς αυτούς. Τρία προκατακτικά σχόλια μπορώ να κάνω. Πρώτον, πιστεύω πραγματικά ότι δεν πρέπει να βιαστούμε. Ως γενική αρχή. Από θεσμικής άποψης σήμερα δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι η Κομισιόν θα υποβάλει νέα πρόταση, ε, ιδιαίτερα αφού βρισκόμαστε και στο τέλος της θητείας της Κομισιόν. Αυτό δεν μπορώ λοιπόν να το κάνω. Τρίτον, πολλά από όσα ακούσατε ε, κινούνται στην καρδιά του προβλήματος. Όπως είπε και ο Πάτρικ και ο Φρανκ, ε, είναι η, απους, η μη πρόσβασή μας ε, σε ε, ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες. Εγώ είπα δεν μπορώ να, δεν μπορώ να πω ότι θα το αναλάβει η Κομισιόν αυτό. Ε, ενδεχομένως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν και η σωστή ακόμη και απονομικής άποψη απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως ακούσατε ομόφωνα εδώ στο πάνελ ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μιλών και είμαστε προβληματισμένοι για το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να βρεθεί κανένα κράτος μέλος σε δυσμενή θέση όσον αφορά την ασφάλεια ή τον ανταγωνισμό. Προσωπικά λοιπόν θα έλεγα ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και αν ε, υπάρχει ε, ε τρόπος να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός τρόπος ε, ε, αξιολόγηση, ε, ευρωπαϊκή αξιολόγηση κινδύνου. Όπως είπε και ο Πάτρικ, υπάρχουν κάποιες δομές συνεργασίας όσον αφορά τις μυστικές υπηρεσίες και τις στρατιωτικές υπηρεσίες. Ενδεχομένως θα μπορούσε μέσα από μια τέτοια συνεργασία να ενισχυθούν διάβλοι επικοινωνίας μια άλλη πιθανότητα που θα μπορούμε να εξετάσουμε είναι να δημιουργήσουμε μηχανισμό αξιολόγησης κινδύνου τρομοκρατικών ενεργειών. Και πάλι, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων είναι ο τρόπος για να αποφύγουμε καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε αυτές τις προοπτικές στο μέλλον. Ο κύριος Παρίνσκι έθεσε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα και να ξανατονίσω ότι όλα τα ζητήματα που κοιτούμε, είτε πρόκειται για το ΣΥΣ του ΚΛΑΣ, όλα αυτά εξακολουθούν να είναι απόλυτη προτεραιότητά μας. Δεν πιστεύω ότι αυτά που έχουν προταθεί στο ΣΕΣ του Plus έχουν κάποια σχέση με αυτό που συζητούμε, αλλά θα το εξετάσω. Επίσης για την ΙΑΣΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή προετοιμασία ενός νέου κανονισμού που θα υποβληθεί του χρόνου. Και παρά το γεγονός ότι κάποιοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις, θα πρέπει να ξανατονίσω ότι η ευθύνη βαρύνει εκείνους που τράβηξαν τη σκανδάλη, εκείνους που εκτόξευσαν τον πύραυλο ή εκείνους που επέτρεψαν σε αυτούς που το έκαναν να το κάνουν και ε, προχωρούμε με τις έρευνές μας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο λόγος για τον οποίο το τόνισε αυτό είναι ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αν ο κακός, ή κακοί είναι αποφασισμένοι να κάνουν το έγκλημά τους, δεν είναι πάντοτε ε, δυνατό να τους αποτρέψουμε. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να το προσπαθήσουμε, αλλά δεν είναι πάντοτε εφικτό να ε, διασφαλίσουμε ότι θα τους αποτρέψουμε. Και από αυτή την άποψη δεν, ο σκοπός μου δεν ήταν να πω ότι δεν είναι δική μας ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά το ποιος και πότε λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρουμε στο ερώτημα που αφορά την ε, British Airways. Εξετάζουμε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά δεν ε, έχω γνώση ότι κάποια, κάποια αεροπορική εταιρεία ή κάποια ομάδα αεροπορικών εταιρεών έλαβαν πληροφορίες για να χαράξουν ε, ένα πιο ασφαλές σχέδιο πτήσης. Αλλά ε, θα συνεχίσουμε να το εξετάζουμε. Επίσης, ε, ρωτήσατε για τις τεχνολογικές εξελίξεις, για το αν ίσως οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην ενισχυμένη ασφάλεια των πτήσεων. είναι ένα πολύ καλό ερώτημα για να δούμε τι θα κάνουμε στο ε, ε, μέλλον. Για την ενημέρωση των επιβιβατών. Αναγνωρίζω ότι κάτι τέτοιο ε, είναι ζήτημα που προβληματίζει τους ε, ανθρώπους, τους πολίτες, αλλά θα πρέπει να, να τονίσουμε και κάποια μειονεκτήματα βλέπουμε, όπως είπε και ο κύριος Ζήλερ, ότι έχουμε ένα νέο είδος συγκρούσεων και δεν ξέρω αν μπορούμε ε, αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε περισσότερες πληροφορίες. Ούτε έχουμε κάποιο μαγικό ραβδί ώστε να καταστήσουμε κάθε πτήση και όλους τους επιβάτες όλων των πτήσεων ασφαλείς. Συμφωνώ και με αυτό που είπε ο Σαλβαντόρε, Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι κάθε Απειλή από τις ε, ε, ρωσικές αρχές να απαγορεύσουν τις υπερπτήσεις είναι απαράδεκτη. Ο λόγος μάλιστα που δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι θα χάσουν πολλά χρήματα. Και αυτό είναι και το, το κεντρικό σημείο της διαμάχης μας με, ε, με τις ρωσικές αρχές. Δεν το έχουν κάνει ακόμα ακριβώς επειδή χρειάζονται τα χρήματα. Κύριε Τιγκράντης, Κάνατε κάποιες παρατηρήσεις για το αν θα έπρεπε ε, η Κομισιόν να ξεκινήσει δική της διερεύνηση των ζητημάτων αυτών. Καταλαβαίνω ότι θα ήταν κάτι τέτοιο ελκυστικό, αλλά πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε επίσημο ρόλο ως Κομισιόν να διερευνούμε δυστυχήματα. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τα κράτη-μέλη. Οι έρευνες στο συγκεκριμένο δυστύχισμα ήταν ταχύτατες. Περιμένουμε τα, προ... τα πορίσματα της έρευνας ώστε να... έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας κάποιες απαντήσεις και ε, να διασφαλίσουμε ότι το πλαίσιο που ορίζεται στο παράρτημα 13 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Αλλά όπως είπα οι ποινικέ έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Και τέλος, να συμφωνήσω με τα σχόλια του Φρανκ Βρένερ... για το τι κάνουμε σε σχέση με το Ισλανδικό ηφαίστειο. Δεν έχει εκραγεί ακόμη, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε προετοιμασμένοι έχει γίνει μεγάλο έργο από τους αερομεταφορείς, από τις αρχές ε, θα εκδοθούν ε, AIP και βεβαίως η Eurocontrol και οι άλλοι οργανισμοί και υπηρεσίε ελπίζουμε να είναι σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με την προηγούμενη έκρηξη του εφαστείου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της συζήτησής μας για αυτό το πολύ δύσκολο θέμα. Βεβαίως πρέπει να εξάγουμε και τα σωστά συμπεράσματα. Ευχαριστώ και τους ομιλητές μας, αλλά και όλους όσοι έθεσαν ερωτήματα. Ελπίζω να απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις, αλλά βεβαίως η συζήτηση συνεχίζεται. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή και μια παγκόσμια λύση για αυτού του είδους τις ε, περιοχές συγκρούσεων. Στη συνέχεια θα, θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα με τον Υπουργό τουρισμού της Ιταλίας.